Uh, Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη του απογεύματο. Ε, να καλωσορίσω τους συναδέλφους που είναι παρόντες. Έχουμε δύο ε, θέματα. Στις 3.30 έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση, ε, όπου θα είναι πρόεδρος ο κ. Παντσέριο, εισηγητής μας, για τα θέματα των ε, γαρωτικών ε, οχημάτων. Και θέλω να καλωσορίσω και τον κύριο David Mayer που ε, είναι υπεύθυνο στο, στο, DG Market, στην ανάλογη μονάδα. Έχουμε μια πολύ σημαντική μελέτη για το βαθμολόγιο ε, συνθήκων καταναλωτή είναι πολύ σημαντική για μας καταναλωτές και αυτή είναι μια ειδική έκδοση. Έχετε εδώ πέρα μια ειδική έκδοση που είναι για το κοινοβούλιο. Είναι μια ειδική λοιπόν έκδοση που θα την και ε, που θα την έχετε για πολλά χρόνια στο μέλλον. Είναι μια ανεπανάληπτη έκδοση ειδικά για μας, την έχουμε μπροστά μας εδώ. Και μετά ε, μπορείτε να μου κάνετε όποια σχόλια, ερωτήσεις θα θέλησετε. Θα σας δώσω τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω όχι μόνο το βαθμολόγιο τους καταναλωτές, αλλά επίσης χθες ε, δημοσίευσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση για ε, την οποία θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε. Όπως είπα, έχουμε δύο ειδών βαθμολόγητα ε, τα οποία είχαμε φέτος. Αυτό που θα σας παρουσιάσω τώρα επικεντρώνεται σε, δύο, σε τρεις πτυχές της ε, νέας αγοράς. Πρώτον, το θέμα των διασυνοριακών, ε, του διασυνοριακού εμπορίου. Πολύ σημαντικό. Δεύτερον, ε, πόσο καλές είναι οι εθνικέ πολιτικές για τον καταναλωτή. καταναλωτικέ πολιτικές μάλλον. Ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα τη εφαρμογή τη νομοθεσίας, οι προσφυγέ και εδώ πέρα εξετάζουμε σε εθνικό επίπεδο θα ήθελα να παρατηρήσετε στο βαθμολόγιο ότι κάθε κάτω μέλος επιμέρους ε, δίνει κάποια επιμέρου σχόλια. Πότε μπορείτε να δείτε στο δεύτερο τμήμα τι γίνεται με το δικό σας ε, κράτος. Λοιπόν, στα δυσανοριακά, το μήνυμα είναι ότι το, το εσωτερικό ηλεκτρονικό εμπόριο πάει μια χαρά, αλλά υπάρχει πρόβλημα με το διασυνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα δείτε, παρατηρήστε στις δύο γραμμές. Η μία είναι σταθερή γραμμή και στην άλλη υπάρχει μια πολύ μικρή άνοδος στο 2009 σε σχέση με το 10 δεν έχει μεγάλη διαφορά. Να παρατηρήσουμε ότι όταν το, αφού το δοκιμάσουν οι καταναλωτές το διασυνοριακό εμπόριο σε αυτήν την περίπτωση, μετά το συνηθίζουν, ε, δεν, δεν έχουν πρόβλημα. Ενώ οι λιανέμποροι από την πλευρά τους ε, έχουν κάποιες αμφιβολίες ακόμα. Μάλιστα μπορούμε να δούμε και μια πτώση. Και θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβολή και από τις δύο πλευρές, και από την προσφορά και από τη ζήτηση. Εδώ είναι παρεόμοια τα στοιχεία στη διαφάνεια, αλλά οι τάσεις. Εδώ όμως ε, βλέπουμε τα άτομα τα οποία έχουν ίντερνετ στο σπίτι τους. Πόσοι από αυτούς ε, ψώνησαν για ε, σωνεριακά από το ίντερνετ. Υπάρχει πολύ ελαφρά άνοδος. Φαίνεται όμως ότι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι εξίσου... Ε, δεν παρουσιάζει περισσότερα προβλήματα σε σχέση με το εσωτερικό ηλεκτρονικό εμπόριο, σε σχέση με τα προβλήματα στις παραλαβές κλπ. Εξετάσαμε το γιατί ε, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. 62% τους ε, φοβούνται ε, κάποια απάτη, ενώ άλλοι για το τι θα Πρόκειται αν δεν υπάρξει μια παραλαβή. Τα θέματα δηλαδή που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας και η επιβολή κυρώσεων όταν κάτι δεν θα πάει καλά για περιπτώσεις απάτης. Έχουμε λοιπόν εντοπίσει, θεωρούμε, τα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Το υπόλοιπο βαθμολόγιο βάζει τα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει το δείκτης συνθήκων για τον καταναλωτή, ένας νέος δείκτης. Ε, οι συνθήκες περιγράφονται ε, στη στρατηγική στη σχετική στρατηγική και στο πλαίσιο για την ανάπτυξη όπως ονομάζεται. Θα μπορείτε να δείτε στο γράφημα στην έκθεση. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με τις συνθήκες για το... τις καταναλωτικές συνθήκες και τι γίνεται με το δίκτυ. Σε κάποιες περιπτώσεις α, υπάρχει άνοδος και μετά πάλι η πτώση. Α, εξετάσαμε το πού ε, σε ποιες χώρες ε, ε, εμπιστεύεται ο καταναλωτής ότι οι αρχές θα εφαρμόσουν την νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων για και διάφορους άλλους δείκτες. Και επίσης για την, τις και τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Υπάρχουν διάφορες. Θα δείτε και διάφορα στοιχεία για, για τα παράπονα που κάνουν οι καταναλωτές στο βαθμολόγιο. Υπάρχουν πάλι μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Και είδαμε και τις οικονομικές συνθήκες των καταναλωτών, κατά πόσον έχουν δει ε, λόγω της κρίσης οι καταναλωτές. Ε, παρατηρήστε το. Υπάρχει μια σύγκριση σε σχέση με το πόσο κατέβηκε το, ε, έπεσε το ΑΕΠ, είναι η MOV ε, το μοβ και το συγκρίνουμε και με την κατανάλωση των οικοκυριών. Σε κάποιες περιπτώσεις ε, μειώθηκε και το εισόδημα και ε, οι, δαπάνε των οικοκυριών. Έτσι λοιπόν οι οικονομικές συνθήκες επηρέασαν ιδιαίτερα τους καταναλωτές. Έτσι θα πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτέ να καλύψουν τις ανάγκες τους σε εποχές που το εισόδημά τους μειώνεται. Η μελέτη που δημοσιεύσαμε χθε ε, πώς να ενδυναμωθεί η θέση του καταναλωτή. Ε, πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν οι αγορές αλλά αυτό που λείπει από το παζλ είναι ποιο είναι ο Ευρωπαίο καταναλωτή, ο μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή. Τι μπορεί να κάνει, τι γνωρίζει. Η Eurostat έκανε αυτή τη μεγάλη μελέτη για να μαζέψει κάποια εμπειρικά δεδομένα, να φτιάξει το πορτρέτο του, του Ευρωπαίου καταναλωτή και πιστεύουμε ότι αυτό το πορτρέτο μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι νομοθέτε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να κατανοήσουμε τι μπορούν να κάνουν καταναλωτές για να σχεδιάσουμε πιο σωστά την ε, πολιτική και θέματα εκπαίδε... ακόμα και εκπαίδευσης. Επιμόρφωση του καταναλωτή. Είδαμε κάποια υποκειμενικά μέτρα, κατά πόσον οι καταναλωτές είναι, έχουν ε, αυτοπεποίθηση, δεξιότητες, επίγνωση. Ακόμα φτάσαμε και στο σημείο να τους εξετάσουμε για τις γνώσεις τους, ας πούμε, για κάποιες σημάνσεις, το κατά πόσο μπορούν να διαβάσουν κάποιες πληροφορίες, να κάνουν κάποιους επιλογισμούς. Οπότε τώρα κατανοούμε καλύτερα πόσο καλοί είναι οι καταναλωτές στο να κάνουν ε, ορισμένε ε, υπολογισμούς, για παράδειγμα, που υποθέτουμε ότι κάνουν. Ένα άλλο θέμα. Ε, προσπαθούμε να βρούμε αν γνωρίζουν ε, τι έχει γίνει για τα δικαιώματά τους, τι, πώς έχει συνεισφέρει σε αυτό το κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε μιλήσει με ανθρώπους, ε, επικοινωνήσαμε και ηλεκτρονικά μαζί τους και υπάρχει και το θέμα το κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να πάνε, φτάσουν σε δικαστήρια, και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι κατανοτές μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και το ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα σε γενικές γραμμές ε, δεν είναι και τόσο θετικά για εμάς που χαράσουμε τις πολιτικές. Οι καταναλωτές δεν είναι τόσο καλά ενημερωμένοι ε, όσο είμαστε εμείς σαν νομοθέτες. Ας δούμε τρία βασικά καταναλωτικά δικαιώματα. Λιγότεροι από τους μισούς γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων σαν που έχουν ως καταναλωτές. Μόνο 28% γνώριζαν ε, για το θέμα της ε, περίοδου χάριτος και όταν υπάρχει πώληση εξ εξεταποστάσεως. Μόνο το 9% ήξεραν για τη... το δικαίωμα τους στην εγγύηση, ότι μπορούν ε, μετά από 18 μήνες να πάρουν ε, πίσω τα λεφτά τους. Και δεν ξέρουν ότι τους καλύπτει η εγγύηση, σύμφωνα με τον νόμο. Και αναγκάζονται και πολλές φορές και ξαναγοράζουν το ίδιο προϊόν. Και εμείς οφείλουμε να, να ενημερώσουμε τους καταναλωτέ και να του βοηθήσουμε να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Και ε, λιγότερο από τους μισού γνώριζαν ότι υπάρχει μια ε, περίοδος ε, που μπορούν να αλλάξουν τη γνώμη του όταν του πουλάει κάτι ένα πλανόδιος, πλασπλασιά. Τώρα, το δείκτη ε, της ενδυνάμωσης, θα λέγαμε, του καταναλωτή σε διάφορες χώρες. Παρουσιάσαμε τα στοιχεία που βρήκαμε στα κράτη-μέλη και θα τα προχωρήσουμε το θέμα μαζί τους. Υπάρχει και ένα έγγραφο εργασίας της Κομισιόν, το οποίο θα σας διανύμεται σήμερα. Και εκεί θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε την επίγνωση του καταναλωτή, ε, την ε, την ενημέρωσή του, την επιμόρφωσή του από τα μέσα ενημέρωσης. Και θα χρειαστεί να θα λάβουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία αυτά. Η μελάτη ήταν μεγάλη και σε εθνικό επίπεδο και αυτό θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία με, το κάθε κράτος μέλος για να κεντρωθούμε στα επιμέρους προβλήματα. Ευχαριστώ. Good. thank you very much indeed, David. I'm sorry. Ευχαριστώ πολύ, David. Λυπούμε που σε στριμώξαμε. Έχουμε πολύ υλικό διαθέσιμο. Και οι συνάδελφοι θα αντλήσουν από αυτό. Και θα το χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Το υλικό. Δημιουργήσαμε μια ομάδα για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο Παμπλαρίας είναι επικεφαλής και ίσως μπορείς να τους επισκεφτείς. Εκεί ίσως συζητήσετε τους δείκτες, τους σαφείς δείκτες που ετοιμάζουν και μπορεί να γίνει δουλειά και για την Επιτροπή μας, πώς θα προσεγγίσουμε διάφορα θέματα ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό προτείνω σαν άμεση αντίδραση. Και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ κάνει δουλειά για τον τομέα λιανικής, το συζητήσαμε το πρωί. Και μπορεί να υπάρξει επαφή και συζήτηση σε αυτό το τομέα. Είναι αργά βέβαια να συμβάλλει σε αυτό, αλλά κάποια θέματα είναι σημαντικά να γνωστοποιηθούν. Έχουμε συγκεκριμένου επιφανεί ε, συναδέλφου. Έχουμε κάποια λεπτά, έχετε κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Μάιερ, ερωτήσεις, ιδέες, πώς να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία του, διότι έχουμε μερικά λεπτά πριν την έναρξη της ακροάσεως. Η κυρία Φένσελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον προηγούμενο μιλητή. Εργάστηκε πολύ καλά. Περιμένω ανυπόμονα την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Η μελέτη είναι σημαντική για τις εργασίες της Επιτροπής μας και για το όλο θέμα, για όλο το χαρτοφυλάκιο. Πρόκειται για κάτι, για ένα έγγραφο πολύ εξαντλητικό, περιέχει πάρα πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία και περιμένω με ανυπομονησία την δυνατότητα να ε, μάθω τι αναφέρεται, να τλήσω μαθήματα. Προκαταρκτικά έχω κάποια σχόλια, θέλω να πω τα εξής. Η στρατηγική της Ευρώπης του 2020 για την ανάπτυξη Εκεί πρέπει να τονιστούν τα δικαιώματα του καταναλωτού. Το κάνουμε εξάλλου. Πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, θα πρέπει να είναι καλύτερα ενημερωμένοι όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Είναι μία από τις προϋποθέσεις για την επιτυχία στρατηγικής για το 2020. Έχω κάποια σχόλια. Τα σχόλια μου αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο. Οι δείκτες αναφέρουν ότι το διασυνοριακό εμπόριο υπάρχει και αναπτύσσεται σε κάποιο βαθμό. Ο καταναλωτής αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Οι διαδικασίες είναι ευκολότερες. Μειώθηκε, χαμήλωσε λοιπόν το όριο, το κατόφλι για το διασυνοριακό εμπόριο. Είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Κάποιες ανησυχίες εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την ασφάλεια που μπορεί να αισθάνεται ο καταναλωτής. Και εδώ έχω κάποια ερωτήματα. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτως ώστε να αποφύγουμε τους φόβους του καταναλωτή που δημιουργούν ε, εμπόδια για μια συναλλαγή διασυνοριακή με ηλεκτρονικό μέσο. Δηλαδή, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι όλος ιδιαίτερος ενήμεροι, να ενημερωθούν καλύτερα. Ερώτημα, πώς, πώς θα το καταφέρουμε αυτό, πώς θα μπορεί ο καταναλωτής να έχει τις αναγκαίες πληροφορίες, να ενημερώνεται καλύτερα. Διότι υπάρχουν Να. Οι καταναλωτές δεν έχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ξέρω ότι πολλοί, πολλοί βουλευτές στην Επιτροπή μας ασχολούνται με το θέμα, προσπαθούν να το λύσουν. Διαβάζοντας λοιπόν αυτούς τους πίνακες, αυτές τις πληροφορίες, ενδεχομένως μπορούμε να βρούμε κάποια λύση, κάποια δράση. Είναι σημαντικό όσον αφορά την ομοθεσία για την εσωτερική αγορά, κάτι που μας απασχολεί και σε σχέση με το λιανεμπόριο. Ξέρω ότι μας λείπει χρόνος, δεν θα χρονοτριβήσω άλλο. Αλλά κλείνοντα θα ήθελα να πω ότι περιμένω ανυπόμονα τη δυνατότητα να απεξεργαστούμε καλύτερα αυτό το ζήτημα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σβέντσεν. Άλλος, στα γρήγορα. David, θες να απαντήσεις. Α, να προσθέσω εγώ κάτι. Χαίρομαι που εξετάσατε και τους παράγοντες ε, του, της προμήθειας εκτός από τη ζήτησης της προσφοράς εκτός από τη ζήτηση. Αναφέρθηκε και η εναρμόνιση των συνοριακών συμβάσεων και η στάση των λιανοπολιτών όσον αφορά αυτό το θέμα. Ίσως χρειάζεται περισσότερη δουλειά να ακολουθήσει. Ας απαντήσετε στο ερώτημα της κυρίας Βένσεν και ίσως ε, θέλετε να κάνετε και κάποια τελευταία σχόλια και θα πάρουμε μαζί μας αυτό το κομψό έγγραφο και θα το μελετήσουμε δεόντως. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από την πλευρά του καταναλωτή, κάποιοι καταναλωτές είναι πολύ ευχαριστημένοι. Χαίρονται να κάνουν διασυνοριακές ε, αγορές και μάλιστα το κάνουν και χαλαρά. Και έχουν εμπιστοσύνη. Και είναι λίγοι αυτοί που ανησυχούν. Περισσότεροι είναι αυτοί που ανησυχούν. Ανησυχούν για τις απάτες, τι γίνεται αν κάτι πάει στραβά, δεν ανησυχούν τα δικαιώματά τους, συμβαίνει στην πράξη αν κάτι πάει στραβά, αυτό τους προβληματίζει. Γι' αυτό να εφαρμόζονται καλύτερα τα μέτρα σε δυσυνοριακό επίπεδο είναι πολύ καλό και αυτό που λείπει ε, για τους ε, καταναλωτές είναι αποτελεσματικός εναλλακτικό ε, μηχανισμός επιλύσεως των διαφορών. Από πλευράς επιχειρήσεων τα πράγματα δεν πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά, ούτως ή άλλως Είδαμε σε μια μελέτη περσινή που κάναμε ότι στι 6 από τι 10 προσπάθειες που έκαναν οι καταναλωτέ να αγοράσουν διασυνοριακά αρνήθηκαν επιχειρήσει να του πουλήσουν διασυνοριακά. Δεν θέλουν να πουλήσουν διασυνοριακά. Και τα στοιχεία από τον πίνακα βαθμολόγηση δείχνουν ότι λιγότερε επιχειρήσει θέλουν να πουλούν διασυνοριακά από ό,τι κατά το παρελθόν. Ευαίσθητη ισορροπία. Δεν έχει νόημα να έχουν πεποίθηση, αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη οι καταναλωτέ και να μην θέλουν να του πουλήσουν διασυνοριακά πρέπει και τι δύο πλευρέ εξίσωση να τι αντιμετωπίσουμε. Είναι δύσκολη η ισορροπία ενδεχομένω. Αν θέλουμε λοιπόν διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, πρέπει να βρούμε λύση και για τι δύο πλευρέ. Ευχαριστώ που το ξεκινήσατε αυτό το θέμα. Θα βασιστούμε από αυτού και είναι καλό να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το έγγραφο, να πάρουν ένα αντίγραφο όλοι οι συνάδελφοι. συνεφώνησε η Επιτροπή ότι θα ετοιμάσουμε μία μελέτη για τις στρατηγικές για τον καταναλωτή, για το μέλλον και είναι πολύ καλό το υλικό που μας δίνεται. Όταν ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας σε αυτό τομέα θα εξετάσουμε το εγγραφό σας, είναι, ήρθε πολύ έγκαιρα και θα μας βοηθήσει. Προσβλέπουμε σε μελλοντική συνεργασία μαζί σας και με τους συναδέλφους σας και σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Καλώς. Uh, περιμένουμε να έρθει ο εισηγητή και μόλις έρθει θα αρχίσει και η ακρόαση. Ήρθε. Uh, Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ να σας καλωσορίσω σε μια ειδική εκδήλωση σήμερα το απόγευμα, που είναι μια δημόσια ακρόαση κατά την οποία θα εξετάσουμε, θα σχολιάσουμε, θα πάρουμε ε, στοιχεία για μια πολύ σημαντική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο για τα γεωργικά και δασικά μηχανήματα, οχήματα και είμαι πολύ ικανοποιημένος που μπορώ να καλωσορίσω τον κύριο Ματίνο που είναι ε, υπεύθυνος του τομέα από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και παρουσίαση και την ε, μελέτη των επιπτώσεων ήταν και το πρωί εδώ. Ακόμα έχουμε πολλά θέματα να εξετάσουμε μαζί. Θέλω να καλωσορίσω και τον Πιέρα Αντώνιο Πανσέρη που είναι ο σκληρά εργαζόμενος εισηγητής μας και σε ένα λεπτό θα του δώσω το λόγο για να παρουσιάσει τα βασικά σημεία που θα μας απασχολήσουν στην ακρόαση. Κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις από μένα. Η ιδέα της ακρόασης είναι να έχουμε όσο γίνεται πληρέστερη ανταλλαγή απόψεων με τους βασικούς εμπλεκομένους εδώ και όπως θα δείτε και από το πρόγραμμα έχουμε βρει αγκάμα ενδιαφερομένων στο θέμα, κατασκευαστές, χρήστες, εργαζόμενοι. Με μεγάλη ε, χαρά καλωσορίζομαι και τους εκπροσώπους των συνδικάτων εδώ γιατί συμμετέχουν πολύ στα θέματα της ασφάλειας αυτού του επαγγελματικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται τόσο πολύ. Και η πρόταση είναι ε, μια επικαιροποίηση και μεταρρύθμιση του κανονισμού για κανόνες κατασκευή στον τομέα αυτό, πολύ σημαντικός τομέας, ένας τομέας όπου είναι πολύ ενεργός παράγων η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές τεχνολογικές εξελίξεις πραγματοποιούνται και χαίρομαι που θα καλωσορίσω και άλλους που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Σε ό,τι μας αφορά, το βασικό θέμα είναι να εξισορροπήσουμε το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς προβλέποντας τις ανάγκες ασφάλειας, λειτουργίας και περιβαλλοντικής προστασίας επίσης σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν τώρα εδώ είναι πρώτα να συζητήσουμε θέματα τεχνολογίας και πώς εξελίσσονται οι τεχνολογίες και τι θα πρέπει να προβλέπει η νομοθεσία γιατί αυτή πρέπει να στηρίζεται, να προσανατολίζεται στο μέλλον και θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για κρίσιμους τομείς ασφάλειας και περιβαλλοντικής απόδοσης, περιβαλλοντικών επιδόσεων. Αυτά θα μας απασχολήσουν και στο φάκελο που πρέπει να έχετε λάβει ερχόμενοι εδώ θα βρείτε στοιχεία για τους ομιλητές, δεν θα τους παρουσιάσω. Θα δείτε λοιπόν το, το βιογραφικό τους, υπάρχουν και αντίγραφα των παρουσιάσεων μετά την εισαγωγή του κυρίου Πανσέρη θα φύγουμε εμεί από εδώ για να μπορείτε ελεύθερα να βλέπετε τις διαφάνειες. Και τέλος θα ζητήσω να σχολιάσουν τα μέλη και οι συγητές και αν έχουμε χρόνο και άλλοι παρατηρητές μπορεί να παρέμβουν ούτε ώστε να υπάρχει διάλογος. Αυτά λοιπόν θα γίνουν τις επόμενες τρεις ώρες. Πρώτα λοιπόν θα καλέσω τον εισηγητή μας να ανοίξει αυτή τη συνεδρία και να μας δώσει τη δική τους προοπτική, να τονίσει κάποια θέματα που θέλει να αναδείξει στην πρώτη συνεδρία. Ο κύριος Παντσέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, στόχος της πρότασης που θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα είναι να θεσπίσουμε εναρμονισμένα ε, διατάξεις και προδιαγραφές για την κατασκευή αυτών των αγροτικών και δασοκομικών οχημάτων, ούτω ώστε να εγγυηθούμε την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερική αγοράς, αν του οράματος υψηλού επίπεδου προστασίας του περιβάλλοντος και της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας και προφανώς να φροντίσουμε και την ασφάλεια των ε, εργαζομένων στον τόπο εργασία. Συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας η πρόταση, διότι απλουστεύει την παρούσα νομοθεσία όσον αφορά την ε, ε, έγκριση των τύπων αυτοκινήτων, βελτιώνει τη διαφάνεια και μειώνει, το διοικητικό άχθος. Αυτή η εισαγωγή είναι μια εισαγωγή ακόμα ανοιχτή και δεν είναι κλειστή και, και μπορώ να δεχτώ ε, αδίποτε προτάσεις βγουν από τη σημερινή δημόσια ακρόαση. Κατά τη διάρκεια διάφορων συναντήσεων με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και με εκπροσώπους της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντοπίσαμε ούτως υπήν ε, διάφορες προσεγγίσεις και διάφορα σημεία που είναι πολύ σημαντικά και θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτά τα σημεία ε, τα οποία θα είναι και αντικείμενο συζητήσεων ε, καθημερινών. Τέσσερις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει ανάγκη συζητήσεων και θα έλεγα και μία συνεισφορά εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων φορέων, ούτω ώστε να συλλεγούν ε, χρήσιμα στοιχεία για την θέσπιση της νομοθεσίας. Αυτά τα σημεία είναι η κατεξουσδότηση πράξης το χρονοδιάγραμμα, η μεταπόληση υπηρεσίες, η ασφάλεια, τεχνικές προδιαγραφές, εκπομπές και τα οχήματα της κατηγορίας U. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, ε, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ η νέα, ε, η νέα διαδικασία για την έγκριση των οχημάτων αυτών ε, είναι κάτι που δημιουργεί κάποια προβλήματα το πότε τεθεί σε ισχύ. Η περίοδος αυτή η προθεσμία, η ημερομηνία το 2014 ε, είναι υπερφορτωμένη νομοθετικά. Και κατεβλήθησαν μεγάλες προσπάθειες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όσον αφορά τη διαδικασία της εγκρίσεως, αδειοδοτήσεως, σε σχέση και με την οδηγία περί εκπομπών, με τους κανονισμούς για ε, τροχοπέδηση κλπ. Και άλλα θέματα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2014 έγινε και το πιστεύουμε αυτό για να μην έχουμε διαφορετικές νομοθετικές πράξεις οι οποίες να αλληλεπιδρούν και να επηρεάζουν μία την άλλη. Και είναι σημαντικό όλα να ενταχθούν σε ένα κανονισμό αντί να έχουμε ένα άθροισμα 20 και περισσότερων ε, απομονωμένων διών. Διερωτώ με μήπως μπορούμε να βρούμε κάποιες ε, λύσεις που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε μια ισορροπία μεταξύ των απαιτήσεων να δημιουργηθούν ε, προδιαγραφές αναρμονισμένες και της ανάγκης ε, που έχουν οι εμπλεκόμενοι φορείς για την έγκριση των οχημάτων. Και να δοθεί μια ανάσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας της πολύ εντατικής για την έγκριση. Λοιπόν, πριν ληφθούν αποφάσεις, πρέπει να αξιολογήσουμε την ανάγκη μιας μεταβατικής περίοδου Ερωτηματικό θέτω εδώ. Θα δούμε ποιε απαντήσει θα είναι δυνατόν να δοθούν σε αυτό το ερωτηματικό, στη δεύτερη πτυχή. Δηλαδή, και τι γίνεται με τη συντήρηση τη υπηρεσία μετά πώληση και, και την ασφάλεια. Όσον αφορά τεχνικά ζητήματα, στο κεφάλαιο 16 που αφορά τι πληροφορίε που χορηγούνται, επί μακρόν ε, αναλύθηκε αυτό το σημείο. Πολλοί υπογράμμισαν την ιδιαιτερότητα που έχει ο τομέα. Υπάρχουν ανοιχτά θέματα όσον αφορά τι συνέπειε θα έχει η νέα πρόταση για τι μεταπόλεις υπηρεσίε και θέματα όσον αφορά την ασφάλεια των καταναλωτών μετά από τι επισκευέ και τη συντήρηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα εγγυήσεων που θα επιτρέψει ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στι απαιτήσει των επιχειρήσεων και σε εκείνε εκείνων που, που κάνουν επισκευέ και πουλούν ανταλλακτικά. Και είναι ανοιχτή συζήτηση και για αυτά τα θέματα ε, και θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα συναθρήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο. Όσον αφορά την ασφάλεια, αυτό είναι θεμελιώδες σημείο και είναι θεμελιώδες για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τη σχέση μεταξύ αυτού του κανονισμού και της οδηγίας της γενικότερης. Βάζοντας από, τα, από την οδηγία τα οχήματα ε, και αυτά τα συγκεκριμένα οχήματα κάποια θέματα που αφορούν ε, την ασφάλεια αυτών των οχημάτων, αν δημιουργήσουμε διαφορά μεταξύ τη οδηγία και τη πρόταση, ίσω δημιουργηθούν κενά. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τι ε, υπηρεσίε του Κοινοβουλίου να κάνει μια μελέτη που ε, κάνει ε, ένα συσχετισμό μεταξύ τη οδηγία για τα οχήματα με αυτήν εδώ την πρόταση όσον αφορά τα προαπαιτούμενα, τα τεχνικά για τι εκπομπέ. Και όσον αφορά το σύστημα τροχοπαίδηση, ε, θέλουμε να προσθέσουμε τι διαδικασίε τι διοικητικέ, όμω αναφέρονται τα συστήματα οχοπαίδησης όπως το ABS, είναι αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση ασφαλείας, αλλά μπορούν να υπάρξουν και άλλοι μηχανισμοί που μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και θα μπορούσαν να αναφερθούν. Και τέλος, όσον αφορά τις κατηγορίες, τα χείρηματα της κατηγορίας U, το ερώτημα αφορά τη συμπερίληψη των κινητών ε, οχημάτων που δεν πηγαίνουν στους δρόμους, εκτός δρόμων, το ότι εντάσσονται σε αυτόν τον κανονισμό δείχνει ότι υπάρχει η ανάγκη ε, να ρυθμιστούν, να καλυφθούν και θέλουμε ε, πάντα να το λαμβάνουμε υπόψη. Δεν μπορούν να ρυθμιστούν ίσως σε αυτό το χώρο, σε αυτό το πλαίσιο. Ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ελκυστήρες ή τροποποιημένα δασοκομικά ε, μηχανήματα στο το παρελθόν. Είναι μηχανήματα που έχουν δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αυτά που συζητάμε. Αυτή η κατηγορία είπαν κάποιοι πρέπει να εξαιρεθεί από τον κανονισμό και θα πρέπει να κατασταθεί από ad hoc κανονισμό. Άλλη λύση θα μπορούσε να είναι να προβλέπετε ένα ειδικό κεφάλαιο που ασχολείται αποκλειστικά με αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία των μηχανημάτων αυτών. Και στο τέλος είναι το θέμα μιας νέας κατηγορίας ε, που πρέπει ε, να δημιουργηθεί T6 ε, δηλαδή τετράτροχα οχήματα που εκτελούν αγροτικές εργασίες εν είδη ελκυστήρων και χρησιμοποιούμε για άλλου λόγους πέραν από αυτούς που να μπορούν να ελκύσουν άλλα μηχανήματα, να τραβήξουν εφορτία για να φτάσουν σε περιοχές που είναι δύσκολο να έχει κανείς πρόσβαση. Μπορούν να θεωρηθούν σαν συμπληρωματικά οχήματα που συμπληρώνουν τη δουλειά που κάνουν τα διάφορα αγροτικά και δασοκομικά ε, οχήματα. Και ακόμα μια άλλη κατηγορία οχήματα που ε, χρησιμοποιούνται για όθηση ή για έλκυση που θα μπορούσαν να μπουν σε ξεχωριστή κατηγορία. Ουσιαστικά, αυτή είναι σύντομη ε, εισαγωγή μου για τη δημόσια ακρόαση, θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και άλλα. Αυτά είναι τα θέματα που θέλουμε να προσφέρουμε σε όλους σας συζήτηση. Στόχος παραγωγική συζήτηση. Να δημιουργήσουμε τον κανονισμό ο οποίος θα ικανοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερου από του εμπλεκομένου φορεί και θα τον υποστηρίζουν οι περισσότεροι. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παντζέρη για αυτήν την ε, εισαγωγή και την πρωτοβουλία για την ακρόαση. Προβάλλεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση και μπορεί να έχουμε και πολύ μεγάλο ακροατήριο που θα ενδιαφέρεται για τις ε, διαβουλεύσεις μας και βεβαίως μπορείτε να μας αποστείλετε και email με τις παρατηρήσεις σας, παρατηρήσεις προς τον κύριο Παντσέρη, κάποιον από τους ομιλητές. Και τώρα θα προχωρήσουμε στις παρουσιάσεις. Θα παρουσιάσω τους ομιλητές σύντομα και μετά τη σειρά και μετά θα ε, πάω στην άκρη. Κάθε ομιλητής θα έχει στη διάθεσή του κατά μέγιστον 10 λεπτά. Έχουμε εξαιρετική τεχνολογία η οποία μπορεί να σας ε, ε, διευκολύνει να παρακολουθείτε το χρόνο σας. Άρα περιμένουμε από σας μεγάλη ακρίβεια. Και εγώ θα πάρω και το σφυράκι μου μήπως και ξεπεράσετε το χρόνο. Θα μιλήσουμε για τεχνολογικές εξελίξεις στα οχήματα αυτά, επιπτώσεις στην ασφάλεια και το περιβάλλον, ο Λάρς Χόλμκβις θα μας μιλήσει πρώτος, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΛΙΠΑ, που είναι η πολύ γνωστή Ευρωπαϊκή Ένωση Προμηθευτών Αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα. Μετά η Σεσίλ Φάβρ, που είναι υπεύθυνη τεχνολογίας και επικοινωνιών για το AECC, που ενδιαφέρονται για τον έλεγχο εκπομπών με καταλήτες. Μαλίο που είναι ε, αντιπρόεδρος της Euromod, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών ε, Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης. Είναι πολύ ειδική στην ε, προμήθεια όλων αυτών και τους εκπροσωπεί ο κ. Ματέη. Ο Χάιριμπερτ Ράιτερ είναι ο πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου της ΣΥΜΑ που κατασκευάζουν γεωργικά μηχανήματα και τέλος ο κύριος Χένρι Κλάιν Βίλιγκαν, ο οποίος εκπροσωπεί την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οχημάτων, κατασκευαστών οχημάτων ε, παντός εδάφους και θα έχουμε μεγάλο πάνελ θα ακούσουμε πολλά ενδιαφέροντα με πρώτο μιλητή τον κύριο Χόλμκβιστ. Μισό λεπτό να απομακρυνθώ για να βλέπω και εγώ τις ωραίες διαφάνειες. Ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή στην ε, κλίπα για όσους δεν τη γνωρίζουν. Η κλίπα δημιουργήθηκε το 59. Σήμερα έχουμε 90 μέλη από τους πιο επιφανείς προμηθευτές και 29 ενώσεις ε, ε, στο εμπόριο. Είμαστε, έχουμε πάνω από 3.000 εταιρείες μέλη και συνεργαζόμεθα κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, ποια είναι η βιομηχανία αυτή αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Έχουμε 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στο βλάδο αυτών στην Ευρώπη. 5 εκατομμύρια από αυτά εργάζονται στα κράτη-μέλη. 1 ε, εκατομμύριο στην αυτοκίνητο, αυτοκινητοβιομηχανία, στους ελκυστήρες, στα φορτηγά και 25 δις ευρώ ε, στην έρευνα και την ανάπτυξη δαπανούν, κατ' κατέτος στον τομέα. Φέτος ε, θα κατασκευάσουμε 18 εκατομμύρια οχήματα στην Ευρώπη και τώρα έχουμε 270 εκατομμύρια οχήματα στο δρόμο με κινητήρες καύσης, ε, και ε, μετά τις πωλήσει. Ε, οι δραστηριότητες μας ανέρχονται σε 100 εκατομμύρια ετησίως. Θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη πρόσβαση, όσο γίνεται μεγαλύτερη αγορά, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε μια ε, εναρμονισμένη παγκοσμίω συνολικά αγορά. Θα ήταν θαυμάσιο αν μπορούσε να επιτευχθεί αυτό, αλλά υπάρχουν συνεχή εμπόδια και προσκόμματα. Κάποια είναι φυσικά, κάποια είναι τεχνητά. Στην Ευρώπη όμως δουλεύουμε μέσα από την ε, Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Ευρώπη στη Γενέβη για αυτό το τομέα που λέγεται Ομάδα Εργασίας 29 και που ασχολείται με παγκόσμιους τεχνικούς κανονισμούς. Καμιά φορά όμως πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά, ε, τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε με μια σειρά, πρέπει να δούμε πώς θα εναρμονίσουμε δηλαδή πρώτα την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη βιομηχανία του κλάδου μας, γιατί αν δεν υπάρχει εναρμονισμένη εγχώρια αγορά, είναι δύσκολο να ανταγωνιστούμε σε, μέσα σε άλλες αγορές. Δύο πράγματα που πάντοτε ήταν πρόβλημα όταν μιλάμε για κανονισμούς είναι η ασφάλεια και το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν είμαστε συνηθισμένοι σε αυστηρότατα πρότυπα ασφαλείας και είναι σημαντικό θεωρούμε να μην λησμονούνται όλα αυτά όταν μιλάμε για το περιβάλλον, για το διοξίδιο του άνθρακα κλπ. Πολλά από τα μέλη μας σήμερα είναι πολύ δραστήρια κατά τη μετάβαση από του παλιού τύπου την παθητική ασφάλεια δηλαδή να γίνονται λιγότερο αισθητά τα αποτελέσματα της σύγκρουσης σε λιγότερο παθητικά, όπου προσπαθείς να αποφύγεις τη σύγκρουση. Αν δούμε όλα τα οχήματα στον δρόμο, πρέπει όλα να είναι ασφαλή, γιατί αλλιώς δεν θα είναι ασφαλές κανένα όχημα στους δρόμους. Πιστεύουμε ότι αυτά τα πρότυπα ασφαλείας που εξετάζουμε σήμερα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα που έχουν άδεια κυκλοφορίας. Εγώ ε, ε, είμαι και λίγο αγρότης, ε, έχω λοιπόν τρακτέρ, τα οδηγώ στους δρόμους, τα είναι, ε, έχουν άδεια και υπάρχουν πολλά, και παλιότεροι ερπιστήρες δηλαδή, καμιά 150.000, ε, πρέπει όμως να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση και οι ίδιοι Τώρα θέλουμε το ABS παντού, θέλουμε επέδυση ε, ταχύτατη παντού, θέλουμε συνεχώς βελτιούμενη ασφάλεια μέσα από πολλά μέσα. Το ABS τώρα είναι 32 ετών αυτό το σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών. Και έχουμε και ηλεκτρονικά συστήματα τα οποία μας βοηθούν σήμερα πάρα πολύ και επίσης είναι ζωτική σημασία γιατί σώζουν ζωές. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο του 50% στη μείωση των θανάτων στους ευρωπαϊκούς δρόμους, θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε όλοι οι εξοπλισμοί να πληρούν τα καλύτερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας. Όταν εξετάζουμε το περιβάλλον, έχουμε την ίδια επιχειρηματολογία. Μιλάμε για το διοξίδιο του άνθρακα για τα αυτοκίνητα, για τα φορτηγά, για τα ελαφρά επιβατηγά οχήματα, μιλάμε για το Euro 6, για τα λεωφορτηγά και τα λεωφορεία και πιστεύω ότι τα, τα αυστηρά αυτά προαπαιτούμενα είναι καλά για τον κλάδο, είναι θετικά για το περιβάλλον, αλλά πολύ δύσκολα ε, ε, πραγματοποιούνται. Ο κλάδος όμως απέδειξε επανειλημμένα ότι προλαβαίνει έγκαιρα να κάνει τα δέοντα, ούτως ώστε τα οχήματα να πληρούν τις προδιαγραφές. Όταν πρόκειται για ε, ελκυστήρες και δασικού εξοπλισμούς, εδώ δεν είναι όπως τα αυτοκίνητα, αλλά μοιάζουν με τα φορτηγά, όπου κατασκευάζονται με κάποια μέρη από τους υπεύθυνου που κάνουν του κατασκευαστές φορτηγών, άλλους που κάνουν άλλου είδους ε, εξαρτήματα. Πολλά προβλήματα έχουμε όταν πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το έργο και το φορτίο που αναλαμβάνουν αυτά τα οχήματα, γιατί δεν είναι μόνο μεγάλα αυτοκίνητα, είναι μηχανήματα που λειτουργούν και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Αλλά έχουμε αποδείξει ξανά και ξανά ότι είναι δυνατόν όλα τα βαρέα οχήματα να είναι αποδεκτά και από άποψη ασφαλείας και από άποψη περιβαλλοντική και είμαστε απόλυτα έτοιμοι να βοηθήσουμε να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Όταν πρόκειται για θέματα επισκευών, συντήρησης είναι σημαντικό να φροντίσουμε, όπως στην αγορά φορτηγών και αυτοκινήτων, ότι θα υπάρχει καλή πρόσβαση στην πληροφορία που χρειάζεται για επισκευές και συντήρηση, ώστε η αγορά να συντηρείται ανοιχτή, ελεύθερη και ανταγωνιστική αγορά. Αυτό έχει ρυθμιστεί ενώ βέβαια έχουμε και το Euro 5, Euro 6 αντίστοιχα για επιβατηγά και βαρέα οχήματα και αυτό είναι καλό παράδειγμα που δείχνει ότι μπορούμε να φροντίσουμε να έχουμε ελεύθερη αγορά. Γιατί σήμερα η μετααγορά aftermarket στην Ευρώπη αποτελείται κατά 50% από επώνυμους dealer και το υπόλοιπο είναι η ελεύθερη αγορά. Εμείς οι προμηθευτές εξαρτημάτων μερών θέλουμε να προμηθεύσουμε οποιοδήποτε που συντηρεί και επισκευάζει αυτά τα οχήματα και είναι καλό το παράδειγμα αυτό ανταγωνιστικής αγοράς όταν υπάρχει πάνω από ένας πελάτης για τα προϊόντα μας. Αυτό που πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την αγορά είναι ότι μαζί με τους ρυθμιστικούς φορείς να συνεργαστούμε. Θέλουμε ρεαλιστικούς στόχους, θέλουμε να φροντίσουμε ότι θα προεξετάσουμε το μέλλον και θα προετοιμαστούμε γι' αυτό. Προς το παρόν βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη, για να μην πω επανάσταση, όταν μιλάμε για επιβατηγά και εμπορικά φορτηγά προκειμένου περί περιβαλλοντικών στόχων. Αν έχουμε ας πούμε τα 120 στα 95 γραμμάρια και όταν αλλάξουμε τον κύκλο δοκιμών και οδήγησης θα πρέπει να φροντίσουμε και θα φροντίσουμε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για να πληρωθούν οι προϋποθέσεις. Το ίδιο θα ισχύσει για όλους τους κινητήρες καύσης που είναι στους δρόμους, γιατί έχουμε το θέμα της ε, θέρμανσης του πλανήτη, της αύξησης της θερμοκρασίας. Ακόμα και για τα δασικά οχήματα, για τα, τους ελκυστήρες θα πρέπει να δούμε το μέλλον και να είμαστε έτοιμοι να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα υγρά κάψιμα γιατί είναι καταλληλότερα για αυτά τα οχήματα, ίσως όμως και τα βιοκαύσιμα. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει και κάποιος εξηλεκτρισμός στην αγορά όπως και στα επιβατηγά, τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Στην βασική μας αγορά επιβατηγών δεν μιλάμε για 10-15 χρόνια από τώρα, αλλά για 2-3 χρόνια. Αυτό είναι ο χρονικός ορίζον όταν θα δούμε την έναρξη του εξηλεκτρισμού. Και σε αυτή την αγορά που, για την οποία μιλάμε μπορεί να απέχει λίγο περισσότερο, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ε, δαπανώνται δισεκατομμύρια ευρώ για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσει του μέλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χόμκουιστ. Δεν είχαμε αντίγραφο από το διαφάνειες να τις εκτυπώσουμε, αλλά θα είναι στην ιστοσελίδα μας, αν τις θελήσουμε. Θα αλλάξουμε τώρα τις διαφάνειες και θα έχουμε άλλη μια παρουσίαση που σχετίζεται με τα σχόλιά σας για τις εκπομπές, δεξιδίου το άνθρακα και τα πρότυπα. Mm. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σιλφάβρ. Mm. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα σας μιλήσω για τις εκπομπές από τρακτέρ και για τα εκτός ε, δρόμου ε, α, εκπροσωπώ το ΑΕΚ. Εδώ πέρα μπορείτε να δείτε διάφορα, τις διάφορες εταιρείες που είναι μέλη μας, που ασχολούνται με ε, τον έλεγχο εκπομπών. Είναι εταιρείε που ε, παράγουν ε, οχήματα εμπορικά και μη, ελαφρά και βαριά οχήματα, μοτοσυκλέτες και off-road εφαρμογές. Αυτή οι εκπομπέ ε, ελέγχονται από την ε, ε, οδηγία που βλέπετε στη διαφάνεια. Το άρθρο είναι σύμφωνο με την οδηγία αυτή, την 9768. Στη τμήμα 3 λέει ότι τα, τα όρια και οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με την οδηγία 97 68. Αν δούμε τώρα α, τη συνολική, συνολική εικόνα πώς την δημοσίευσε η Κομισιόν, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπομπών είναι από τον α, εκτός δρόμου κλάδο μηχανημάτων. Μπορούμε να το δούμε στο 2005, το 2010 και το 2020 τα ποσοστά. Παρόλο που το ποσοστό μειώνεται, όμως ε, οι αγροτικές εφαρμογές είναι ε, μέχρι και 50% αντιπροσωπεύουν στο κάτω μέρος της διαφάνειας. Η συνολική μείωση δεν είναι τόσο μεγάλη όπως πριν και παραμένει μεγάλο το ποσοστό των αγροτικών εκπομπών. Είναι σημαντικό οι εκπομπές από τρακτέρ να συνεχίσουν να, είναι, να υποκείται σε κανονισμούς και στην νομοθεσία. Τώρα για τα όρια εκπομπών. Το 2013 το πιο αυστηρό στάδιο, το στάδιο 4, ε, πλησιάζει αυτά που είναι και στην κάτω, στο κάτω γράφημα. Πολλοί κατασκευαστές έχουν διαφημίσει πρωτότυπα για μηχανές σε στάδιο 4 που δεν θα έχουν τα φίλτρα για τα διοξίδια του αζότου. Στην επόμενη διαφάνεια η Επιστημονική Ένωση, η κάναμε πέρσι ένα πρόγραμμα δοκιμαστικό, το οποίο εξελίχθηκε για το στάδιο 3B. Δεν θα σας πω πολλές τεχνικές λεπτομέρειες. Βασικά, να σας πω με λίγα δεν υπήρχε πρόγραμμα ελέγχου των εκπομπών χρησιμοποίησαμε ένα σύστημα calibration Ένα πλήρες σύστημα ελέγχου εκπομπών ε, μας το παρέχει το ΑΕΚ. Περιλαμβάνει το, τον έλεγχο του σωματιδίου. Το σύστημα εδώ πέρα μπορεί τον, της, εξα, ε, είναι το μήκος το οποίο είναι κλασικό στις βιομηχανικές ε, στα βιομηχανικά μηχανήματα. Τώρα, στις επόμενες διαφάνειες, θα με τις εκπομπές που έχουν μετρηθεί. Ε, υπάρχουν διάφοροι κύκλοι κύκλοι δοκιμών. Οι κόκκινες γραμμές είναι τα, τα όρια του, του σταδίου 4, το πιο αυστηρό όπως είπαμε προηγουμένως. Πέρα από αυτές τις πολύ χαμελές εκπομπές, το σύστημα ε, ελέγχεται Α, θα το περάσουμε στην επόμενη εκπομπή που αφορά τα εκπομπέ εξοδίων του αζότου. Η μεταβολή είναι πολύ, με... η... είναι πολύ μεγάλη στις περισσότερες ε, κύκλους δοκιμών, στους περισσότερους κύκλους δοκιμών. Τα όρια του 2-4 είναι... γίνονται σεβαστά, με κάποια εξαίρεση. και η μεταβολή των οξυδίων του αζότου ως αποδοτικότητα εξαρτάται από την θερμοκρασία. Μετά η, η μείωση των εκπομπών σωματιδίων είναι μέσα στα όρια, με μεγάλο περιθώριο. Και η αποδοτικότητα είναι μεταξύ 60-67% στους κύκλους που αναφέρονται. Τώρα για τη μελλοντική νομοθεσία. Μπορούμε να δούμε τα ποσοστά των σωματιδίων. στο γραφείο μου. Ε, βλέπουμε λοιπόν είναι 10 στην 11η κάτω από 9 μικρότερο το 9 μικρότερο από το 10% χιλιόγραμμα ένα κιλοβατόρο. Ε, η συνδυασμός σύγχρονου συστήματος μηχανής με ένα σύστημα ελέγχου εκπομπών ε, οδηγήσαμε σημαντικές μειώσεις σε όλα τα ελεγχόμενα σωματίδια και σε όλους τους ελεγχόμενους ε, μολυντές και τις ελεγχόμενες πηγές μόλυνσης. Τέλος, να πω σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι εκπομπές ε, από τα δασικά και ε, αγροτικά μηχανήματα θα συνεχίσουν να, να αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό των συνολικών εκτός δρόμου εκπομπών, σωματιδίων και διοξιδίων του αζότου. Πρέπει να, να, υπάρξει, να συνεχιστεί αυτή η ευθυγράμμιση με την ε, νομοθεσία για τον εκτός δρόμου οχήματα όχι μόνο στο στάδιο 4 αλλά και παρα, παρα, παραπέρα. Καλό θα ήταν να υπάρξει εισαγωγή ενός αριθμού, ενός ε, σωματιδίων και θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας ένα μελλοντικό στάδιο 5. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Well, thank you very much for... Um, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε όλοι να παρακολουθήσουμε τις λεπτομέρειες. Uh, Από τα διαγράμματα μετά θα καταλάβουμε καλύτερα και κάποια θέματα που θίξατε θα συζητήσουμε αργότερα. Αυτή είναι η γενική έποψη εκείνων που ετοιμάζουν εξοπλισμό με βάση τους καταλήτες. Τι γίνεται με τους κατασκευαστές των κινητήρων, οι οποίοι εγκαθίσταται δεν εγκαθίστανται σε αυτό το υλικό. Ο κύριος Ματέι έχει αυτό το θέμα, θα μας μιλήσει γι' αυτό. Καταρχάς, ευχαριστώ εκ μέρου τη ενώσεω μου που μα καλέσατε να συμβάλλουμε στη συζήτηση. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την εισαγωγή που κάνατε. Αυτό είναι το Euromod. Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση των κατασκευαστών, Ευρωπαίων Κατασκευαστών Κινητήρων Σωτερικής Καύσεως. Είμαστε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των κατασκευαστών των κινητήρων εσωτερική καύση που παρέχουν του κινητήρε στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω Υποστηρίζαμε τα μέλη μας από το 1991 ε, δίνοντας τους τεχνογνωσία και ενημερωμένες πληροφορίες και κάνοντας εξαρτήσεις εκ μέρους τους για διεθνώς ευθυγραμμισμένη νομοθεσία. Είναι φορέας ευρωπαϊκών συμφερόντων η Euromod και είμαστε στο μητρό διαφάνειας με τον αριθμό που βλέπετε εκεί. Αυτό είναι ο αριθμός μητρό μας. Ε, συλλέγουμε μάλλον περιλαμβάνουμε και όχι μόνο στην Ευρώπη, 40 κατασκευαστές ε, κινητήρων, 40 εταιρείε από την μικρότερη μέχρι την πολυεθνική καλύπτουμε. Τα μέλη της Euromod, δηλαδή τι θέλουμε να κάνουμε όσον αφορά την ποιότητα. Θεωρούμε ότι τα μέλη της Euromod θέλουν να λάβουν μέτρα αποτελεσματικά όσον αφορά το κόστος για να βελτιώσουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζονται στην ολοκλήρωση προϊόντων για το στάδιο 4 των κινητών των, της οδηγίας 1997-68 ε, ΕΟΚ για τις εκπομπές μηχανημάτων εκτός δρόμου και θέλουμε να συμβάλλουμε στις συζητήσεις για την επόμενη φάση ε, των απαιτήσεων για εκπομπές αυτών των οχημάτων, στάδιο 5, κάνοντας μια μελέτη κόστος ωφέλους ε, και αξιολόγηση συνεπιών για την ε, κοινωνία. Να υπενθυμίσω ότι από την αξιολόγηση αντιχτύπου του GRC το 2007 ο εξοπλισμός εκτός δρόμου συμβάλλει 9% σε εκπομπές σωματιδίων στην Ευρώπη και αν περιορίσουμε αυτή την συνεισφορά στα κάτι μέλη, τα 15 κάτι μέλη, είμαστε μόνο στα 5%, όμως θέλουμε να συμβάλλουν συζητήσεις για το στάδιο 5 όσον αφορά τον καθορισμό ορίων εκπομπών των οχημάτων εκτός δρόμου. Ποια θέματα θέλω να υπογραμμίσω. Η έγκριση της οδηγίας NRMM, της οδηγίας 9768, για ελκυστήρε αγροτικού και δασοκομικού, ενημέρωση τη οδηγία 97-68 και συνέπειε για τη γεωργία και για του ελκυστήρε του γεωργικού και του δασοκομικού τομέα, τη θέση ισχύ του κανονισμού και ποιε είναι οι απαιτήσει OBD. Η οδηγία 9768. Η Euromod καλωσορίζει την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε μία και μόνο οδηγία που καθορίζει την απέτηση για τους, τα μηχανήματα αυτά, τα NRMM και τους ελκυστήρες. Οι προθεσμίες εφαρμογή σήμερα είναι ταυτόσιμες αλλά έχουν διαφορετικό νόημα. Για τα NRMM, δηλαδή τα μηχανήματα εκτός δρόμου και τη σχετική οδηγία, η, η ημερομηνία καθορίζει ότι η ημερομηνία επιτίθεται το όχημα στην αγορά, ενώ η οδηγία 2025 για τους ελκυστήρε συμπίπτει με τη θέση υπηρεσία του ελκυστήρα. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Υπάρχει διαφορά ημερομηνιών και η διαφορά αυτή είναι το ελάχιστο έξι μήνες στην πράξη. Όλες οι ημερομηνίε ε, ισχύω για τους ελκυστήρες έχουν έρθει πιο κοντά, είναι πιο πρώιμοι συγκριτικά με τους NRMM, τουλάχιστον κατά ένα εξάμεινο. Πριν η Euromod, γι' αυτό προτείνουμε με την υιοθέτηση της 9768 για τους ελκυστήρες να ευθυγραμμιστεί η προθεσμία και για την ε, τοποθέτηση των ε, κινητήρων στην αγορά. Όσον αφορά την αλλαγή της νομοθεσίας, την εξέλιξη της νομοθεσίας για τις εκπομπές, οδηγία 9768, αυτή αναθεωρείται πλήρως. Θα ισχύει είτε άμεσα στους ελκυστήρες ή μέσω των μεταφορών της οδηγίας 2025. Θεωρούμε ότι το θέμα που συζητούμε αποτελεί τμήμα της αναθεώρησης της 68 και παρόλα αυτά γίνεται ε, μία ανάλυση συνεπιών για να επικαιροποιηθεί η οδηγία 2025 ΕΟΚ. Η ημερομηνία υλοποίησης εφαρμογής. Ο κανονισμός προτείνεται να εφαρμοστεί από 1η Πρώτου 2007 είχε προταθεί. Όμως Απάμε, αυτό αφορούσε και τι, τι γίνεται από την, το να περάσουμε από τη φάση 3β μέχρι 4. Είναι θέμα το να απολυθούν ε, τα αποθέματα και οι σχετικές διατάξεις για την πόλη των αποθεμάτων θα έχουν σοβαρές συνέπειες. Γι' αυτό ζητάμε η υποθεσμία θέση ισχύ να καθυστερήσει τουλάχιστον 1η Πρώτου 2017, ζητώ συγγνώμη, ζητά συγγνώμη διερμηνία, όχι 2007, 2017. Ε, και αυτό να ταιριάξει με την εφαρμογή της οδηγίας για τα NRMM. Ε, τα χρώματα στο διάγραμμα βλέπετε την, ε, δείχνουν την, την προθεσμία, την ημερομηνία εισαγωγής του μέτρου και πώς σταδιακά εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες. Μεταβατικά στάδια. Από 1η Πρώτου 2014 θα εισάγουμε, θα δούμε θα πάμε 75 με 130 στην ισχύ. Και κάποιο που θέλει να δοθεί πιστοποιητικό σε νέο ελκυστήρα με τον νέο κανονισμό θα ζητήσει κινητήρα στα 2-4 πάνω από ένα χρόνο πριν τη θέση ισχύ του 97-68. Και οι ρήτρες περιπολίσεως διετίας θα καταργηθεί από 130 μέχρι 360 κιλοβατόρες ο κανονισμός για αυτά τα οχήματα καταργεί την προθεσμία διετών για την πώληση του αποθέματος. Αυτό υπονομεύει τη βιομηχανική δυνατότητα που θα έχει ο τομέας όσον αφορά τη σταδιακή εισαγωγή νέων προϊόντων και σταδιακή ε, εξάλληψη των παλαιών. Απαιτήσει OBD, κεφάλαιο 16 του κανονισμού. ο κανονισμός για, τις, ε, για τα οχήματα δρόμου δεν καλύπτει την περίπτωσή μας. Θέλουμε να μην υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει παρέμβαση στα οχήματα για να μην ξεπεραστούν ε, τα διάφορα όρια. Υπάρχει σχετική διάταξη που θα εμποδίσει τη λειτουργία του ελκυστήρα αν το σύστημα ελέγχου της εξάτμισης δεν λειτουργεί σωστά. Το BD λοιπόν, ένυψη, ελήψη ε, τακτικών ελέγχων είναι αδύναμο εργαλείο για τις εκπομπές. Και σχετικό λογισμικό, OBD, θα ανοίξει το, το δρόμο σε hacking, κόλπα. Και άρα θα πετύχουμε τα, τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Γι' αυτό Euromod ζητά η αναφορά στο OBD να καθυστερήσει, να μην ακολουθηθεί Υποθεσμία. Και το λογισμικό που ελέγχει τους κινητήρες θα πρέπει να φυλάσσεται από παρέμβαση, από hacking με άλλα λόγια. Λοιπόν, πώ συνοψίζουμε την πρότασή μας. Αυτά τα τρία πράγματα προτείνουμε. Η Euromod υποστηρίζει την, την υιοθέτηση της οδηγίας 9768 ΕΟΚ για γεωργικά τρακτέρ υπό τον όρο ότι η ημερομηνία θέση ισχύ θα είναι η ίδια και για τα τρακτέρ και για τα άλλα οχήματα εκτός δρόμου και τα μηχανήματα. Ζητάει η Euromod η ημερομηνία θέση ισχύ του κανονισμού να καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι 1ου 1ου 2017. Η Euromod ζητά η αναφορά στο OBD να διαγραφεί από το κεφάλαιο 16. Ευχαριστώ. Right. Well, thank you very much. I think we'll clearly return. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αναφερθήκατε και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει λιγάκι στις ερωτήσεις θα αναφερθούμε σε κάποιες τεχνολογίες και σημεία επαφής οχημάτων εκτός δρόμου και τα διαγνωστικά συστήματα μέσα στο αυτοκίνητο και τις ναι. προτάσεις για τα γεωργικά μηχανήματα. Ναι. Μην ναι. χρησιμοποιείτε πολύ ακρονίμια γιατί δεν τα ξέρουν όλοι. Ε, λοιπόν, ο κύριος Ράιτερ θα μας μιλήσει τώρα ε, από την ε, ΣΕΜΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να παρουσιάσω τη ΣΥΜΑ που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που εκπροσωπεί τα γεωργικά μηχανήματα στην Ευρώπη εδώ και 50 χρόνια και καλύπτει πολυεθνικές μέχρι χιλιάδες μικρομεσαίες με ένα ισχυρό ε, δίκτυο 10 εθνικών οργανώσεων μελών που αναγνωρίζεται ως εταίρος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Επόμενο παρακαλώ. Ο κλάδος ε, πίσω από την ΣΕΜΑ, 4.500 κατασκευαστές, 21 δις ευρώ παραγωγή, στοιχεία του 2010, 250.000 απασχολούμενοι 135.000, άμεση απασχολούμενοι 125 πρόσθετοι στο, στη διανομή και στο σέρβις. Καλύπτουμε 400, 450 ε, διαφορετικά μηχανήματα, τρακτέρ, ε, σταθερά, πρόσθετα, συνδυασμένα, ε, μηχανήματα, συγκομιδής κλπ. Τώρα, τρία βασικά θέματα. Το ένα είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεύτερον, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κινητά μηχανήματα και πώς θα απλουστεύσουμε τα μηχανήματα ε, σε σχέση με τις ε, ε, επιδόσεις τους. Ε, βλέπετε εδώ το άρθρο 64 που είναι βάση. Αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος ε, έχει χρόνο για να έχει ετοιμάσει όλες τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Δεν υπάρχει σταδιακή εισαγωγή νέων τύπων ε, μηχανημάτων με τον τρόπο που αυτό διασφαλίζεται από την οδηγία και ο κλάδος είναι στο μέσο μιας δύσκολης διαδικασίας εγκρίσεων για το στάδιο 4 κυρίως που θα πρέπει να ολοκληρωθεί 1η Ιανουαρίου του 2014 όπως ακούσαμε ε, στα 130 κιλοβάτα και 1η Σεπτεμβρίου του 2014 για την υποδύναμη πιο κάτω. Η πρόταση θα είναι ότι η θέση σε ισχύ δεν θα είναι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της τελευταίας κατεξουσιοδότηση πράξης που είναι απαραίτητη για όλη την έγκριση, ολόκληρη την έγκριση του τύπου οχήματο ε, και των κατηγοριών μετά την τελευταία εισαγω... Ε, ημερομηνία εισαγωγή ε, του προγράμματο εκπομπών και λαμβάνοντα υπόψη δύο χρόνια προσαρμογή στι διοικητικέ αλλαγέ 2015 συν 2 λοιπόν. Κάποιος χρόνος χρειάζεται για την προετοιμασία διοικητικών αλλαγών και πιθανές τεχνικές αλλαγές όπως την πέδηση που θα εφαρμοστούν την περίοδο μέχρι το 2014. Επίσης το 2014 θα υπάρξει μια μεγάλη σύγκρουση στη βιομηχανία γιατί θα πρέπει καταρχήν να έχουμε το, τις εκπομπές που θα πρέπει να ε, πληρούνται οι προδιαγραφές και μετά θα πρέπει να έχουμε ένα νέο πλαίσιο. Το επόμενο θέμα, κάποιες ευθυγραμμίσεις και απλουστεύσεις στον τομέα. Ο στόχος του κανονισμού είναι να ευθυγραμμίσουμε τις διαδικασίες έγκρισης τύπου όλων των τομέων υπό την ε, επίβλεψη της μονάδας της Κομισιόν για τα αυτοκίνητα. Το άλλο είναι να γίνει η αναρμόνιση και απλούστευση για τους στόχους αυτούς. Ε, η πρόταση της ΕΜΑΣΕΣΕ είναι η κατηγορία 2 να εξαιρεθεί από την, το μητρικό κανονισμό και το δεύτερο είναι να απλουστεύσουμε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ως προς τις πρόσθετες ε, υποκατηγορίες. Θα σας δείξω τι εννοώ αργότερα με ένα slide. Τώρα για τους, για τα, τους ελκυστήρες έχουμε την έγκριση του τύπου, ε, στον κανονισμό τον αρχικό η αξιολόγηση επικινδυνότητας γίνεται από εμπειρογνώμονες και έχουμε τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην νομοθεσία και η, ε, ο ε, σεβασμός στα πρότυπα ελέγχεται με, από τις αρχές έγκρισης τύπου μετά για την αυτοταυτοποίηση ε, γίνεται από τον κατασκευαστή η αξιολόγηση επικίνδυνοτητας, εναρμονισμένα πρότυπα για να βοηθήσουν ε, ε, στην εφαρμογή, δήλωση αξιοπιστίας από τον ίδιο, εποπτεία αγοράς που ελέγχει. Επίσης, έχουμε σήμερα τους τρεις πυλώνες επαγγελματική ασφάλεια περιβαλλοντική προστασία οδική ασφάλεια και στην ε, δήλωση από τον ίδιο καλύπτεται από την οδηγία για τα μηχανήματα ή επαγγελματική ασφάλεια και από την οδηγία για το θόρυβο και τις εκπομπές η περιβαλλοντική. Η οδική ασφάλεια δεν έχει ακόμη εναρμονιστεί. Τώρα, ε, μηχανήματα εκτός δρόμου, ε, αν μπουν στο νέο κανονισμό, τότε θα πρέπει τα μηχανήματα να ε, καλύπτονται από το πλαίσιο των κανονισμών και πρέπει να πληρούν την αυτοπιστοποίηση ε, για την ε, επαγγελματική ασφάλεια και περιβαλλοντική προστασία και θα πρέπει με την οδική ασφάλεια να ακολουθούν τον μητρικό αρχικό κανονισμό. Επόμενο. Τώρα, γιατί η προσθήκη της κατηγορίας U στην, ε, στο μητρικό κανονισμό δεν είναι ενδεδειγμένη. Έχουμε δύο σειρές ε, νομοθεσίας ε, που θα δημιουργούσαν σύγχυση και διοικητική επιβάρυνση. Τα μηχανήματα κατηγορίας U εμπίπτουν στον νέο κανονισμό με βάση τη νέα προσέγγιση, οδηγία για τα μηχανήματα και όλα τα θέματα ασφάλειας εκτός από την οδική. τι θα γίνει με τις διπλής χρήσης μηχανήματα. Ε, τεχνικές προδιαγραφές ε, για τις, τα κινητά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τις κατασκευές είναι πιο κοντά, προσεγγίζουν μεταξύ τους πιο πολύ από ότι ε, οι ελκυστήρες και τα κινητά γεωργικά μηχανήματα. Επίση, αν είναι προαιρετική η κατηγορία U, τότε δεν θα χρησιμοποιείται και δεν θα ισχύουν οι προδιαγραφές. Λόγω της υψηλή ποικιλομορφία των οχημάτων κατηγορία U, θα καθυστερούσε η ε, πρόοδος του κανονισμού. Ε, τώρα, μηχανήματα εκτός δρόμου, έχουμε τον τύπο, την έγκριση τύπου, έχουμε και την αυτοπιστοποίηση. Ε, η οδική ασφάλεια θα αντιμετωπίζεται μέσα από το, την οδηγία για τα μηχανήματα, είναι ο κανονισμό, τα άλλα δύο θα καλύπτονται από τις οδηγίες ε, εκπομπών και θορύβου και θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των ε, μηχανημάτων αυτών. Επίσης προτάσεις ευθυγράμμισης και απλούστευσης για τους ελκυστήρες. Τώρα έχουμε κάτω από 40 χιλιόμετρα και τώρα έχουμε ε, για μεγαλύτερη υψηλότερη ταχύτητα και προβλέπουμε και άλλη κατηγορία. Η πρότασή μας στην επόμενη διαφάνεια είναι η εφαρμογή υποκατηγοριών α και β ενώ η κατηγορία Α θα καλύπτει ελκυστήρες κάτω από 40 χιλιόμετρα, ενώ το Β άνω των 40 χιλιόμετρων και το 1Β για παράδειγμα θα αντικαταστήσει την κατηγορία ΤΑΦ5. Το πλεονέκτημα και ο λόγος για την πρόταση αυτή είναι, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, να αποφύγουμε απειλές από πιθανές νέες κατηγορίες στο μέλλον θα έχουμε μία απλούστευση του πεδίου εφαρμογής με υποκατηγορίες και θα έχουμε λιγότερες κατηγορίες. Επίσης, η ταχύτητα χρήση ειδικών προϋποθέσεων για την διεύθυνση, υπέδηση κλπ. Όλες οι άλλες οι προϋποθέσεις θα είναι ίδιες για τις υποκατηγορίες. Η καταλληλότητα της πρότασης είναι ότι δεν χρειάζεται ε, ταχεία κατηγορία τρακτέρ TAF5. Η διαγραφή του TAF5 θα πρέπει να συνδέεται αυστηρά με τη δημιουργία υποκατηγοριών Α και Β και αυτές είναι προϋποθέσεις για τρακτέρ με ταχύτητα άνω 40 χιλιόμετρων. Η δυνατότητα υπάρχει, αν λάβουμε υπόψη μας την υψηλότερη ταχύτητα και έτσι θα έχουμε ένα θετικό μήνυμα προς τα έξω. Επίσης θα υπάρχουν δυνατότητες ε, ε, καινούργιοι για τους κατασκευαστές ελκυστήρων. Τα προαπαιτούμενα κριτήρια και ορισμοί θα πρέπει να είναι ε, ακριβείς ε, προκειμένου να καλυφθούν νέα οχήματα που μπαίνουν στον κανονισμό γεωργικών οχημάτων. Συνοψίζω, η πρόταση κανονισμού για τα προβλήματα σχετικά με τα γεωργικά οχήματα, απλούστευση διαδικασιών έγκρισης τύπου, μείωση διοικητικής επιβάρυνσης, ευθυγράμμιση με τους κανόνες για τα αυτοκίνητα. Η βιομηχανία συμφωνεί με τα περισσότερα, όμως το κεφάλαιο 16, πρόσβαση στην επισκευή των οχημάτων, αυτό θα το αναφέρει άλλος ομιλητής και το χρονοδιάγραμμα πρέπει να ε, προσαρμοστεί για να έχουν χρόνο. Οι προτάσει τη ΣΕΜΑ για την ευθυγράμμιση και την απλούστευση απλουστεύουμε το πεδίο εφαρμογή και ε, ορθολογικοποιώντας το για τις κατηγορίες, με τις κατηγορίες ΤΑΦ, ΑΒ, υποκατηγορίες και αφαίρεση της κατηγορία U ε, και εναρμόνιση της οδικής ασφάλειας και των προδιαγραφών για το κινητό μηχανισμό οδικό κανονισμό που θα ευθυγραμμίζεται με τις ε, οδηγίες νέου νομοθετικού πλαισίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν μας διευκολύνεται, αλλά θα είναι πολλά θέματα τα οποία ανέκυψαν δεν είναι μόνο η μελλοντική τεχνολογία που θέλαμε να ακούσουμε από εσά, αλλά και διάφορα νομοθετικά ζητήματα. Αλλά για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τόσο καλά τη δουλειά μας, γιατί είχαμε δουλέψει στην οδηγία για τα χανήματα και τον εξοπλισμό, εμείς τα γνωρίζουμε καλύτερα. Κάποια θέματα που ανέκυψαν τότε. Και εδώ και πολύ καιρό ζητάμε αυτή την οδηγία για τα τρακτέρ αλλά πολλά θέματα για, θέματα που υπάρχουν, υπάρχουν υπερκαλύψεις για τα εκτό δρόμου μηχανήματα και οχήματα. Τα καλύψει ο πιο μετά ο εισηγητής. Ας περάσουμε τώρα στην τελευταία παρουσίαση της, του, του, του τμήματος. Νομίζω ότι ο κύριος Βαν Βίλιγκελ θα μας μιλήσει. Νομίζω ότι έχετε και εσείς κάποιες υπόψεις για την συμπερίληψη με κάποιων κατηγοριών οχημάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε μπροστά στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σα πω ποια είναι η ΑΤΒΕΑ. Είναι η Ένωση των Ευρωπαϊκών της, ε, βιομηχανίας των οχημάτων ε, για όλα τα εδάφη. Ε, έχουμε, παραγωγή ψυχική ε, παραγωγή 100.000 ε, μονάδες το χρόνο περίπου, είναι μυστικά μικρή, που καλύπτεται από τις εταιρείε της ΑΤΒΕΑ. Όμως είναι πολύ ε, ε αγαπητά οχήματα στους Ευρωπαίους χρήστες. Ε, και αντιπροσωπεύουμε το 67% των συνολικών πωλήσεων χημάτων ΑΤΒΕΑ, τύπου ΑΤΒΕΑ. Το υπόλοιπο καλύπτεται από 40 με 50 κινέζικες εταιρείε. Έχουμε προσπαθήσει να του ε, κάνουμε μέλη στην ενωσή μα, αλλά χωρίς επιτυχία, διότι φαίνεται ότι δεν του ενδιαφέρει και τόσο με τέτοια συμμετοχή. Το πεδίο εφαρμογή ε, το εύρο τη ΑΤΒΕΑ ε, είναι για οχήματα που βασικά ε, έχουν σχεδιαστεί για μη ασφαλτοστρωμένε επιφάνειες. Αριστερά βλέπετε κλασικά off-road οχήματα. Δεξιά μπορείτε να δείτε κάποια άλλα τύπου οχήματο, που να έχουν τις μάρκες των μελών μας στο ντεπόζιτο, αλλά είναι με πειραγμένα θα λέγαμε οχήματα που έρχονται προσφορές από εκτός Ευρώπης είναι, έχουν χαρακτηριστικά τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν τη δική μας α, ε, ενώση. Εμείς ε, ε, ιδρυθήκαμε για να ενημερώσουμε τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις αρχές ε, για αυτά τα τίποτα οχήματα. Νιώσαμε την ανάγκη να ενημερώσουμε το κοινό ορθά. Τώρα αυτά, αυτά τα επαγγελματικά ATV και SBS side by side, πώς γίνεται η έγκριση τύπου σήμερα. Ε, δεν υπήρχε στην Ευρώπη κάποια ξεκάθαρος ορισμός, ένας ξεκάθαρος ορισμός για αυτό το τύπο τα οχήματα, τόσο από την Ισπανία και την Πορτογαλία όπου έχουν, ε, κάνει έχουν δημιουργήσει ένα είδο έγκριση τύπου για αυτά τα προϊόντα. Οπότε βασικά τα προϊόντα μα ε, ε, λαμβάνουν την έγκριση τύπου ε, σαν τρακτέρ στη Γερμανία, με επίσης μια νομοθεσία ευρωπαϊκή, πολύ λίγο θα έλεγα, ad hoc σε, κάποιες, σε κάποια και είναι και το, η έγκριση L6 και 7 που αφορά τα, τα μικροαυτοκίνητα, γουρούνες και, τα ETV καλύπτονται από αυτό το έγκριση τύπου. Τα ETV είναι ε, για, όλες, για όλα τα ίδια έχουν σχεδιαστεί γι' αυτό και αυτό το κάνει το, το πιο την εγκρισιτή τύπου πιο παρήπλοκη, ακριβώς γι' αυτόν λόγο. Αλλά ε, αυτά τα, ε, οι συνομοθεσίες δεν καλύπτουν επαρκώς το πεδίο. Γι' αυτό και ζητάμε να υπάρξει ένα σωστό νομικό πλαίσιο για τα, με την, στον κανονισμό για τα αγρο, αγροτικά και δασικά οχήματα, για τα επαγγελματικά ATV τα επαγγελματικά ATV είναι μια κατηγορία των ATV. Και πιστεύουμε ότι η σωστή κατηγορία είναι τα αγροτικ... η κατηγορία των αγροτικών και δασικών οχημάτων. Εκεί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περιβαλλοντικά και ε, ζητήματα και τα ζητήματα ασφάλειας με το καλύτερο τρόπο. Τώρα για τα οχήματα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των επαγγελματικών ATV και SBS είναι πάντα μικρά και ελαφρα. Γι' αυτό έχουν και μικρή κατανάλωση καυσίμων και έχουν και μικρότερες εκπομπές δεξιδίου το άνθρακα. Είναι αρκετά οικονομικά σε σχέση με άλλα επαγγελματικά οχήματα που χρησιμοποιούνται σε αγροτικό και δασικό περιβάλλον και έχουν επίσης τη μεγάλη δυνατότητα να, έχουν πρόσβαση σε διάφορα τύποι εδαφών που δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερα οχήματα. Και είναι και πολύ ωραία ο τρόπος που συνδυάζονται μαζί με τα τρακτέρ. Έχουν μια συμπληρωματικότητα. Μιλήσαμε για τα side by side και τα ATV. E Μπορεί να αναρωτιόσαστε ποιες είναι οι διαφορές τους κάποια χαρακτηριστικά. Τα, τα επαγγελματικά ETV έχουν ε, ένα δικό τύπο α, σέλας που μοιάζει με τις μοτοσυκλέτας. Ε, ο οδηγό πρέπει να μπορεί να κινείται πάνω στη σέλα δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω για να μπορέσει να έχει καλύτερη πρόσβαση στο έδαφος αν φτάσει σε κάποιο λοφίσκο, χρησιμοποιεί το βάρος του για να ξεσορροπήσει. Έχει επίσης ε, κάποιο ειδικό ε, τιμόνι θα λέγαμε. Ε, υπήρχε όμως ζήτηση για κάποια πιο σταθερά οχήματα σε, να σε αυτό το περιβάλλον και γι' αυτό ε, το side by side. Εδώ ο οδηγός είναι δίπλα, κάθεται. Έχουμε ένα παραδοσιακό τιμόνι. Ε, είναι πιο ψηλό το, το όχημα σε σχέση με άλλα σχετικά και υπάρχει και η δυνατότητα ρημούλκησης. Και το κάθισμα είναι παραδοσιακό. Ε, χρειάζεται μεγάλες δυνατότητες μεγαλύτερη ισχύ και σχέση με το έδαφος. Τώρα, μπορούμε να δούμε εδώ τη διασύνδεση με την οδηγία για το τακτέρ. Μπορούμε να δούμε αριστερά τα... Ε, τα χαρακτηριστικά, όπως αναφέρονται στο κάθε περιοχή, κάθε κομμάτι της νομοθεσίας. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η σωστή νομοθεσία είναι αυτή που μας αφορά ο κανονισμός τεταρκτέρ. Γιατί είναι απαραίτητα οχήματα αυτά τα ATV e και τα SBS για την δασοκομεία και την, ε, τις αγροτικές εργασίες. Είναι σχεδιασμένα για ακραίες συνθήκες δαφικές. Έχουν μικρό ε, αποτύπωμα ενεργειακό περιβαλλοντικό θα λέγαμε. Ε, είναι μια οικονομική λύση για συγκεκριμένες εργασίες ε, στο, σε αγροτικό περιβάλλον. Παλιά οι Άγγλοι αγρότες έπρεπε να κυνηγούσαν τα πεζή τα πρόβατα, τώρα μπορούν να το κάνουν πάνω σε αυτά τα οχήματα. Επίσης υπάρχουν ε, πολύ ψηλά πρότυπα ασφάλειας τα οποία είναι σύμφωνα με την ε, οδηγία για, τους, για τα μηχανήματα. Τώρα, οι, ε, οι εμπλεκόμενοι για την ΑΤΒΕΑ είχαμε μια συνεργασία στο παρελθόν με την Γενική Διεύθυνση για τις ε, Enterprise, την επιχειρηματικότητα, από το 2004, στα πλαίσια της αναθεώρησης των πλησίων TKL. Πρόσφατα πήγαμε και σε εμπειρογνώμενα σε κάθε κράτος μέλος και σε ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μάθουμε τις απόψεις τους για τέτοιου τύπου οχήματος, οχημάτων και είδαμε ότι υπάρχει ένα όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτά τα οχήματα και άρα και για την νομοθεσία που είναι σχετική. Χρειάζεται βέβαια μία ξεκάθαρη, ξεκάθαρης ορισμός για να ξεχωρίσουμε αυτά τα επαγγελματικά ε, οχήματα από άλλα οχήματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία L. Τα συμπεράσματα για να βελτιωθεί η κατάσταση θα ζητήσουμε από τις αρχές να να υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών που προκύπτουν από τη χρήση των συγκεκριμένων οχημάτων. Θα θέλαμε να συζητήσουμε να, περιλαμβάν, να περιλάβετε τα ITV και τα SBS στην, στο νέο πλαίσιο, κανονιστικό πλαίσιο T, TAF. Επίσης, χρειάζεται προετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών στα κατεξοδίου της πράξης, με βάση τη σωστή κατηγοριοποίηση των οχημάτων και η Ατβέα τέλος είναι πάρα πολύ ανοιχτή ε, σε ανταλλαγή απόψεων μαζί σας, να σας δώσουμε κάθε πληροφορία που θα χρειαστείτε. Γιατί πιστεύω ότι η τεχνονοσία αυτού του προϊόντος δεν είναι και τόσο ευρέως δεδομένη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας άφησα να μιλήσετε περισσότερο, διότι δεν είναι πολύ συχνά που έρχεται κόσμο κόσμος και μας ζητά να θεσπιστή ρύθμιση για να τους πλησιώσει. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι ο εισηγητής μας για τα οχήματα τύπου L, ο κ. Βαντενκάμπ είναι εδώ και ασχολήθηκε με κάποια από τα άλλα θέματα που αναφέρατε ε, και με τα οχήματα επιδρόμου. Πάνε παράλληλα οι δύο προτάσεις βλέπετε για τα διάφορα ίδια οχήματων. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα είναι εύκολο, αλλά ίσω θα πρέπει να καλέσουμε του συναδέλφους να υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις, να διερευνήσουμε κάποια από αυτά τα θέματα και σε κάποια φάση ίσως ζητήσαμε από καθέναν από εσά να συνοψίσετε τα βασικά σας σημεία. Τώρα για τα στοιχεία φωτισμού και το side by side καινούριο είναι αυτό που ε, καινούριο όρος που άκουσα και για τον ελαφρύ εξοπλισμό επίσης που αναφέρατε. Προτείνει κάποιες εξαιρέσεις από την πρόταση του Dr. Ράιτερ. κάποιοι θέλουν να μπουν μέσα, κάποιοι να βγουν έξω, μπορεί να τα συζητήσουμε. Και αλληλεπικάλυψη μεταξύ των κατηγοριοποίησεως εκπομπών οχημάτων εκτός δρόμου και τι γίνεται με τα οχήματα δρόμου και κάποιοι είπαν ότι χρειάζεται κάποια ευθυγράμμιση. Υπάρχουν μηχανικοί που χρησιμοποιούν τους ίδιους κινητήρες σε κατηγορίες μηχανημάτων, σε διαφορετικές κατηγορίες μηχανημάτων. Δεν έχει νόημα να σας ζητούν οι ρυθμιστικές αρχές να μια δουλειά δύο φορές. Μπορεί να το διερευνήσουμε το θέμα. Περιμένουμε νέες τεχνολογίες, νέες εξελίξεις. Ξέρουμε κάποιες νέες τεχνολογίες. Μας ανέφερε η βιομηχανία κατασκευής καταλυτών. Ε, θα πρέπει κάποια από τα θέματα να τα συζητήσουμε. Και πότε θα τοποθετηθούν αυτά τα εξαρτήματα. Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουν οι ερωτήσεις, ξεκινώντας από τον κύριο Βαντερ Κάμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν είμαι σκιώδης εισηγητής για τους, για τους ελκυστήρες, αλλά είμαι εισηγητής για την έγκριση τύπου των οχημάτων κατηγορίας L. Τους περασμένους μήνες μιλήσαμε με την ΕΔΕΑ αρκετές φορές, όμως μετά την παρουσίαση έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, η αναψυχή θεωρείται κάτι και κάτι σαν εργαλείο η αναψυχή θεωρείται ένα όχημα αναψυχής μπορεί να θεωρηθεί και επαγγελματικό όχημα ταυτόχρονα που κάνει κάποια δουλειά. Ε, γίνονται πολλές συζητήσεις. Υπάρχουν πολλά οχήματα επαγγελματικά βαριά και side by side οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αναψυχή, για διασκέδαση. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουν σε άλλες χώρες, όπως τις είπα. Λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει η διάκριση μεταξύ των χρήσιμων μηχανημάτων, των επαγγελματικών και των μηχανημάτων και των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για αναψυχία. Υπάρχει και άλλη κατηγορία ίσως οχημάτων που, οχημάτων σας που στην κατηγορία L. Θέλετε όλα τα οχήματα παντός εδάφους να μπουν εκεί. είχατε διαγράψει αυτά τα οχήματα. Δεν θα καλύπτονται καθόλου ή θα μπουν στην κατηγορία L. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Μετά, ξέρουμε ότι κάποια οχήματα από αυτά χρησιμοποιούνται και επί δρόμου. Δεν ξέρουμε αν είναι νόμιμο ή όχι, δεν το συζητάμε αυτό. Θα έπρεπε η αστυνομία να κάνει κάτι γι' αυτό, να επιβάλλει τον νόμο. Ας υποθέσουμε ότι έχει ένα όχημα με πλάγια θέση side by side και αυτό βγαίνει στο αυτοκινητόδρομο. Ποια νομοθεσία ισχύει για αυτή η περίπτωση. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που έχω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάιλερ έχει το λόγο. Εγώ δεν θα μιλήσω για τεχνικά θέματα. Κάποιος ομιλητής αναφέρθηκε στη χρονική στιγμή θέση σε ισχύ της οδηγίας και ποια είναι η καλύτερη στιγμή και πολλοί εξέφρασαν την επιθυμία να αναβληθεί η τη. Πριν από 7 χρόνια συνεργάστηκα για την οδηγία για τα μηχανήματα και στη συζήτηση τότε σκοπίμως τους ελκυστήρες τους είχαμε αφήσει απ' έξω και η βιομηχανία το ήθελε αυτό γιατί προφανώς είπαν ότι οι προϋποθέσεις για την οδηγία για τα μηχανήματα δεν μπορεί να ταυτίζεται με εκείνη για τους ελκυστήρες. Θα κάνουμε δικό μας. Το καταλάβαμε, το θεωρήσαμε σωστό. Τότε, πριν από 7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν απόλυτα σαφές για όλους τους συμμετασχόντες ότι θα υπήρχε κάποια στιγμή μια οδηγία για τους ελκυστήρες. Πολύ συγκεκριμένα, ειδικά για αυτό τον κλάδο με αυτή τη στόχευση δηλαδή ελκυστήρας. Στους ελκυστήρες όλοι θα μπορούσαν να ξέρουν ή θα έπρεπε να ξέρουν ότι κάτι θα γινόταν. Γι' αυτό με εκπλήσει λίγο που θέλετε κι άλλη αναβολή στο χρονοδιάγραμμα της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Κι εγώ για το ίδιο να πω κάτι. Οι πρώτοι δύο ομιλητές, η ομιλήτρια και ο ομιλητής, οι δύο πρώτοι, είπαν σαφώς ότι οι τεχνικές προδιαγραφές υφίστανται για να τεθούν αυτές οι απαιτήσει, ενώ η βιομηχανία λέει ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Δεν το καταλαβαίνω. Υπάρχει η ίδια αντίφαση που είχαμε ε, μεταξύ των δύο. Η βιομηχανία θέλει πιο πολύ χρόνο, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι και εμείς αντιμετωπίζουμε πιέσεις. Έχουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής, το είπατε, και γι' αυτό νομίζω ότι δεν γίνεται να αναβάλουμε κι άλλο. Αν οι κινητήρες και στα λεωφορεία μπορούν να ε, τοποθετούνται όπως στους ελκυστήρες, τότε οι διαφορές δεν είναι πολύ μεγάλες. Από την άλλη, μπορούμε να τηρούμε λοιπόν τις προδιαγραφές και κατά δεύτερον το ότι χρειάζεται ακόμα ας πούμε, μια περίοδος 2-3 ετών ε, είναι πολύ, δεν το καταλαβαίνω γιατί τόσο. Άλλος συνάδελφος που θέλει να πει κάτι, ο κ. Μάντερς. Δύο πράγματα. Συμπληρώνω καταρχάς το ερώτημα του φίλου μου, του Ρενέ Βαντερκάμπ. Αν αυτά τα οχήματα πάνε στο δημόσιο δρόμο υπάρχουν οι ίδιες απαιτήσει ασφαλείας. Χρειάζεται ειδική αδειοδήγηση. Και για τα δίτροχα οχήματα. Είναι σημαντική η ορατότητα, αλλά και για τα γεωργικά. Και το θέμα του φωτισμού που αναφέρατε ε, επίσης παίζει ρόλο. Σαν νομικός έλεγα, όπου υπάρχουν εξαιρέσεις, δημιουργεί σφαιά νομική ζώνη. Θα ήταν δυνατόν ίσως να αποφύγουμε τις ε, εξαιρέσεις. Υπό την ιδιότητα του σκιώδου συζητητού του κυρίου Παντζέρη και όχι του Πρόεδρου να πω κάποια πράγματα. Αυτό που είπε η κυρία Βάιλερ για την ελεπικάλυψη με την οδηγία για, το, για τα διάφορα μηχανήματα. καταλαβαίνουμε πού υπάρχει το σημείο επαφή μεταξύ των δύο ρυθμίσεων. Κύριε Ράιτερ, μας δείξατε ένα διάγραμμα χρωματιστό. Ειδικέ απαιτήσει ασφαλεία για οχήματα μπορούν να βγουν στον δρόμο σε κάποια φάση. Αλλά το όχημα αυτό ουσιαστικά είναι εξοπλισμός. Μπορεί να είναι γεωργικός εξοπλισμός, ε, εξοπλισμό για κατασκευέ κλπ. Τι γίνεται όταν βγει στον δρόμο. Υπάρχουν διαφορέ στι εθνικές νομοθεσίες για τις απαιτήσει όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Όλοι συμφωνούν και η Ένωση Κατασκευαστών αυτού του εξοπλισμού μας είπαν ότι όλα τα μέτρα πρέπει να εναρμονιστούν. Έκανε κάποιες προτάσεις οι κατασκευαστές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εναρμόνιση. Θέσατε το ερώτημα, χρειάζεται νέο κανονισμό είπατε, αν, αντί να υπάρχει κατηγορία you λατινικό, να βρεθεί τρόπο εναρμόνισης των απαιτήσεων ασφαλείας για εξοπλισμό που ίσως μπορεί να βγει και στον δρόμο και χρησιμοποιηθεί στον δρόμο, αλλά ε, κατασκευή είναι εξοπλισμός, μηχάνημα. Έναντι άλλου υλικού που μπορεί να ταξινομηθεί ως ελκυστήρας. Έχω δίκιο? Γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο αυτό που άκουσα. Δεύτερον, τρακτέρ που τρέχουν πιο γρήγορα και αλλαγέ στην κατηγορία 5. Αναφέρατε κάποιε τι αλλαγέ. Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε ξέρω για αυτά τα τρακτέρ που τρέχουν. Αρκετά μίλια έκανα πρόσφατα σε τέτοιο τρακτέρ, όμως σε τέτοιο τρακτέρ. Χτύπησε 50 χιλιόμετρα την ώρα το τρακτέρ ασφαλέστατο, άνετο, ήσυχο ήταν. Και οι κατασκευαστές αυτού του μηχανήματος θέλουν να εγκριθεί. Το επιθυμούν διακαώς. Τέτοιου είδους τρακτέρ υψηλής ταχύτητας, πού εντάσσονται κατά άποψή σα, Από ό,τι κατάλαβα για κάθε κατηγορία, τρακτέρ, μεγέθου τρακτέρ, από ένα μέχρι τέσσερα θα έχετε τις ισχύουσες προδιαγραφές και υποκατηγορία για τρακτέρ που κινούνται πιο γρήγορα. Θα έχουν IBS, προχωρημένο σύστημα τροχοπαίδησης κλπ. Θα προβλέπετε αυτό. Περί αυτού πρόκειται, αυτό αναφέρατε. Και τα τρακτέρ που υπάρχουν σήμερα πάνε πιο γρήγορα βάσει τη προτάσεώ σα. Μπορούν να εγκριθούν πλήρω και να πάρουν έγκριση τύπου οχήματο. Δεν τα ξεκάθαρο. Αυτά έχω να πω αρχικά, ίσως να έχουμε χρόνο και για άλλο γύρο ερωτήσεων. Θα καλέσω τους ομιλητές σε αντίστροφη σειρά να αναφερθούν στα σημεία. Για τον Dr. Ράιτερ και τον κύριο Βαν Βάλεγκεν και τον κύριο Ματέι είναι τα βασικά τα περισσότερα ερωτήματα, αλλά λέει ασχολιάσουν και άλλοι, ο κύριος Βαν Βίνεγκεν για να αναφερθεί στα ερωτήματα του κυρίου Βάντεν Κάμπ για το θέμα της αλληλεπικάλυψης. Για τα ελαφρά τρακτέρ, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσετε αυτά ή τα side by side. Νέες λέξεις, νέα, νέα ορολογία για σήμερα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Εμείς μιλάμε για η βίας με φέλη μου φορτίου, να το πούμε επαγγελματικά, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και όσο οχήματα αναψυχής, αν το θέλει κανείς, μόνο που δεν είναι και τόσο όμορφα. Η Ατβέα είπε, όλα τα μέλη δηλαδή είπαν, ότι σίγουρα πρέπει να έχουμε ATV, ωφέλη μου φορτίου, στην γεωργική οδηγία. Κάποιοι ψάχνουν ακόμα δυνατότητες να έχουμε και αναψυχή ε, με βάση την παλιά οδηγία. Αν τα ETV χρησιμοποιούνται και για σκοπούς αναψυχής, πρωτίστως θα γίνεται αυτό εκτός δρόμου συνθήκες εκτός δρόμου που μοιάζουν με τις συνθήκες λειτουργίας και τις τεχνικές προδιαγραφές των ελκυστήρων. Γι' αυτό το συζητάμε ακόμα το θέμα. Όταν μιλάμε για αναψυχή, έχουμε δύο έννοιες εδώ. Το ένα είναι ο αθλητισμός και τα σπόρο οχήματα που μπορούν να χρησιμοποιούνται ιδιωτικά και ε, με τους τύπους των σπόροχημάτων που χρησιμοποιούνται στο δρόμο με ημιτροποποιημένες εκδοχές. Αυτά δεν θα συνεχιστούν για αυτά τα μοντέλα για λόγους ασφαλείας. Αυτό το έχουμε δεχτεί. Ελπίζω ότι απάντησα επαρκώς. Είχα και μια συμπληρωματική, αλλά μπορεί και εσείς να κάνατε την ίδια. Πείτε λοιπόν. Δεν ξέρω. Αν λέτε ότι χρησιμοποιούνται τα εκτός δρόμου ως σπορ, πού θα πάνε στην κατηγορία L ή TAF. Όχι στην TAF, σίγουρα όχι για τα σπορ και για κάποια από τα... Έχουμε την κατηγορία για τα τετράτροχα ε, εκτός δρόμου. Όχι για εν, ε, εντός δρόμου ε, χρήση. Αυτό θα πρέπει να καλύπτεται ε, στα 15, στις Γι' αυτό μιλάμε για τον κανονισμό των ε, ΤΑΦ. Ο Δόκτωρ Ράιτερ. Για το χρονοδιάγραμμα με ρωτήσατε για την ε, εφαρμογή, τη θέση σε ισχύ. Η βασική τεχνολογία είναι στη διάθεσή μας, αλλά βλέπουμε αλλαγές στο σχεδιασμό. Στα 2, 3 και 4 είναι σημαντικές, θα αλλάξει όλο το μπροστινό. Για τους ε, ελκυστήρες, για τον κινητήρα, ο βασικός κινητήρας είναι ο ίδιος στα λεωφορεία και τα φορτηγά, αλλά απ' την άλλη η εγκατάσταση κάθε μηχανήματος είναι διαφορετική και πρέπει να γίνονται προσαρμογές στο περιβάλλον αυτό για τα τρακτέρ, είναι μεγάλη τροχή. Θα πρέπει επίσης να δούμε τι είναι το σύστημα διεύθυνσης και όλα αυτά. Επίσης, πρέπει να κάνουμε όλες τις αλλαγές στα σχέδια, πολύ βραχυπρόθεσμα και πρέπει να εγκαταστήσουμε μεγάλα μέρη στα τρακτέρ, για παράδειγμα, και ειδικά μηχανήματα που που συχνά δεν υπάρχει χώρος για την εγκατάσταση. Γι' αυτό εμείς στην εταιρεία μου δαπανούμε πάνω από το 70% των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης στις αλλαγές των σχεδιασμών για να ανταποκριθούμε στις προδιαγραφές εκπομπών. Επίσης θέλουμε να ε, εγκαθιστούμε τους κινητήρες νωρίτερα, κάνοντας όμως όλες τις μεγάλες αλλαγές στα σχέδια. Αυτό είναι πρόκληση για τον κλάδο των προμηθευτών γιατί τα συστήματα ε, ε, εκπομπών και σέρίων έχουν ε, διαφοροποίησεις. Δεν είναι τυποποιημένα τα μέρη, πρέπει να έχουν ειδικό σχεδιασμό για να ταιριάζουν στους εξοπλισμούς τους δικούς μας. Ε, σας έκανα και άλλες δύο ερωτήσεις, αν μπορείτε να απαντήσετε για τις προδιαγραφές ασφαλείας και για την πρότασή σας κατάργησης του ΤΑΦ5 και α, για την ε, διαγραφή του ΤΑΦ5 αν υπάρχει προσθήκη υποκατηγορίας δεν χρειάζεται πρόσθετη κατηγορία τρακτέρ θα υπάρχει μια σειρά κατηγοριών και αν ο τρακτέρ είναι ταχύτερος από 40 χιλιόμετρα τότε θα πρέπει να έχουμε ειδική εκδοχή B και ειδική διαδικασία έγκρισης τύπου. Αυτό απλουστεύει τη συνολική διαδικασία έγκρισης τύπου. Και το, η άλλη ερώτηση ήταν για τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές οδικής ασφάλειας για οδικούς εξοπλισμούς. Τώρα οι προϋποθέσεις για την οδική ασφάλεια δεν είναι εναρμονισμένες και θέλουμε ένα πλαίσιο για την εναρμονισμένο πλαίσιο και να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ έγκριση τύπου και την αυτοπιστοποίηση για τις, τον οδικό εξοπλισμό. Αν η οδική ασφάλεια μπορεί να εφαρμόζεται επίσης σε αυτό το πλαίσιο της εκτός δρόμου, ε, των εκτός δρόμου με ε, ειδικό πλαίσιο ή με αυτοπιστοποίηση για τα μηχανήματα, ώστε η διαδικασία έγκρισης τύπου για τα τρακτέρ και ε, για τους εξοπλισμούς εκτός δρόμου να είναι ανεξάρτητες. Προβλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο παράρτημα για τις ε, οδικές προδιαγραφές ε, που θα εφαρμόζεται και στην οδηγία για τους εξοπλισμούς, γιατί από τι είδα από τους κατασκευαστές εδώ και ένα χρόνο είχαν βάλει τέτοιες προδιαγραφές και είχαν, τις είχαν καταθέσει και στην Κομισιόν. Το έχετε δει αυτό. Ναι, αυτά τα παραρτήματα θα πρέπει να είναι σημεία αναφοράς ή έγγραφα αναφοράς. Άλλοι συνάδελφοι μπορούν να παρέμβουν σχετικά με αυτά που είπαμε για τις δυσκολίες εγκατάστασης, τοποθέτησης των νέων καταλητικών συστημάτων που μας ε, τα παρουσιάσατε τόσο ωραία, γιατί είναι περιορισμένος ο χώρος του ελκυστήρα και του κινητήρα του ελκυστήρα και είναι δύσκολο μηχανολογικά να γίνει η εγκατάσταση. Και ίσως θα πρέπει να γίνει και ε, χωριστή δοκιμή γιατί τα συστήματα εξάτμισης έχουν ειδικά χαρακτηριστικά κάθε φορά. Ίσως λοιπόν μπορείτε να μας πείτε εσείς οι δύο για αυτά. Ε, ίσως δεν ε, θα δώσω την απάντηση που περιμένετε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν, πολλές πρόσθε... υπάρχουν πολλοί πρόσθετοι περιορισμοί στις εφαρμογές μας και προσπαθούμε να τα καταφέρουμε. Όπως είπε ο συνάδελφος ο κύριος Ράιτερ, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι πραγματικοί για να απαντήσω στην κυρία Ρούλερ, δεν μιλάμε για καθυστέρηση χάρη στις ε, συσκευές αυτές ε, της μετά από την ε, κατασκευή. 97-68 έχει σαφή οδικό χάρτη μέχρι το στάδιο 4. Έχουμε δύο after treatments, όπως είπε και η κυρία Φαύρε. έχουμε για τα σωματίδια και έχουμε και μετέπειτα επεξεργασία για τα όρια. Ζητάμε καθυστέρηση, αναβολή, όχι για λόγους τεχνικούς έχουμε και εμείς υιοθετήσει τα ίδια τεχνικά μέτρα καταπολέμησης που θα έχει και στο μέλλον και η Euro 5 και η Euro 6, αλλά το μόνο είναι ότι ο κανονισμός αυτός αλλάζει το νομικό πλαίσιο του ε, τωρινού κανονισμού. Δεν έχει να κάνει με εκπομπές, δεν έχει να κάνει με τεχνική ε, βιωσιμότητα και σκοπιμότητα, αλλά βιομηχανική σκοπιμότητα διότι ακόμα δεν έχουμε όλες τις ε, ε, τροποποιήσεις ε, για το στάδιο 4 και είναι δύσκολο να το εφαρμόσουμε. Η επαγωγή δεν έχει ακόμα ξεκαθαριστεί και μιλάμε και για νέο κανονισμό που θα έρθει σε μία περίοδο όπου η βιομηχανία θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί από οικονομική άποψη και ο κανονισμός θα καταργούσε την έγκριση τύπου την καινούρια ή την διάταξη για τις ε, πωλήσει. Δεν είναι θέμα λοιπόν τεχνικό, δεν έχει να κάνει με τα σωματίδια, τις εκπομπές, ε, ε, δεν έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή είναι θέμα επιχειρησιακό, αν θέλετε. Ε, ναι, και από την άλλη πλευρά, όπως εξήγησε και ο κύριος Ράιτερ, θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στην αγορά. Καμιά φορά λοιπόν πρέπει να γίνεται αξιολόγηση με βάση μελέτη επιπτώσεων, διότι αν δεν προσφέρουμε ε, υψηλών επιδόσεων εξοπλισμούς, λειτουργικούς, που θα αντιστοιχούν τουλάχιστον στους παλιούς, μπορεί να παρατηρηθεί μείωση της αντικατάσταση του παλιού, των παλιών μηχανισμάτων στην αγορά και αυτό θα επηρεάσει τη συνολική ποιότητα. Γιατί στους εξοπλισμούς του δρόμου δεν έχουμε πολιτική ε, διάλυσης των παλιών. Υπάρχουν 30 χρόνων εξοπλισμοί που κυκλοφορούν και έτσι οι εκπομπές είναι πολύ υψηλές. Οπότε πρέπει να τεχεί αυτό το ζήτημα. Πάντως δεν πρόκειται τώρα περί αυτού. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Η κυρία Φάβρα. Να προσπαθήσω να δώσω κάποια ικανοποιητική απάντηση στην ACC δεν θεωρούμε, δεν εξετάζουμε σε ελκυστήρες αυτού, κάθε αυτούς. Υπάρχουν περιορισμοί για τους ελκυστήρες όπως και για τα άλλα οδικά μηχανήματα εξασφάλιση εξασφάλισης του οδηγού, προστασίας του οδηγού και άλλα δύσκολα θέματα αλλά υπάρχουν καλές μηχανολογικές πρακτικές γενικά να τονίσω αυτό που είπα στην παρουσίασή μου. Κάποιοι κατασκευαστές διαφήμισαν μηχανήματα κατηγορίας 4 που δεν θα έχουν φίλτρα για σωματίδια από κινητήρες δίζελ. Άρα ίσως χρειαστεί νέος σχεδιασμός, δεν ξέρω αν ε, χρειάζεται να γίνει νέος σχεδιασμός για τέτοιου είδους φίλτρα για το στάδιο 4. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι να πω, μάθαμε πώς να λύνουμε τα περισσότερα προβλήματα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Πώς όλα αυτά τα συσκευέ και αυτά που απαιτούνται να τα βολέψεις μέσα στο σύγχρονο αυτοκίνητο, στο σύγχρονο ελκυστήρα. Ο Δόκτωρ Ράιτερ είπε ότι 70% έρευνα και ανάπτυξης ε, τα διαθέτει τα ποσά αυτά για τις εκπομπές. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ο κ. Ματίνα είναι εδώ, άκουγε πολύ προσεκτικά. Πολλά αναφέρθηκαν. Σχολιάστε τώρα και παρεμβαίνετε και στο επόμενο στάδιο. Ίσως πάρετε κάποιο χρόνο που σας έδινα μετά, τώρα, αλλά θα ήταν καλό να ακούσουμε την άποψή σας. Σύντομα όμως σας παρακαλώ. κάντε τετράλεπτο σας βολεύει, αν μπορείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα και πάλι στους, στα μέλη τη ΕΜΚΟ που ήταν το πρωί για ένα άλλο θέμα. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσουμε σαν κομισιόν. σίγουρα αυτή η πρόταση είναι πολύ σημαντική για μας. Και αν μου επιτρέπετε, να πάρω μία από τις ε, λέξεις της εισαγωγής σας. Να, θα μπορούσε να είναι οδηγό για τα σχόλιά μας. Οπότε η λέξη κλειδί και η πρόκληση είναι... Λοιπόν, ο κράτος του τρακτέρ έχει ε, υποφέρει από μια διάσπαρτη νομοθετική προσέγγιση, διάσπαρτες νόμους. Ε, Πρόσφαση η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό πεδίο δεν είναι πλήρης και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εκλογικεύσουμε, να απλοποιήσουμε και προσεκτικά να σχεδιάσουμε τις απαιτήσει, τις προδιαγραφές στην νομοθεσία, ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο του, της νομοθεσίας στον κλάδο. Από την άλλη, πρέπει να εκλογικεύσουμε το συνολικά το σύστημα έγκρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω αυτό, εκφράστηκε στις παρουσιάσεις, οπότε για μας ενώ αναγνωρίζουμε τις ε, ε, ότι είναι ειδική κατηγορία τρακτέρ, πρέπει συνολικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να υπάρχει μια συνοχή. Το πρόβλημα τώρα της, ε, το, της, χρόνου. Ε, έχουμε προσπαθήσει και στο παρελθόν ε, με το θέμα των αυτοκινήτων. Αυτοί που τώρα εξετάζουν την κατηγορία L γνωρίζουν ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα συγχρονισμού. Ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όποτε αποφασιστεί να γίνει εφαρμογή, να τεθεί σε ισχύ νομοθεσία, θα πρέπει να έχουμε ένα σωστό πακέτο, το οποίο θα είναι πολύ απλό στην εφαρμογή του, πολύ ξεκάθαρο και το χρονοδιάγραμμα είναι μέσω μακροπρόθεσμο. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν υπόψη και όλες τις τεχνολογικές εξέλιξεις, ώστε να μπορεί να είναι σε εφαρμογή για πολλά χρόνια η νομοθεσία. Ε, είμαι λίγο φυλακτικός για κάποια επιχειρήματα που λένε ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις ε, σε σχέση με την υπάρχουσα νομοθεσία που θα, θα τεθεί σε ίσχυ. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν α, σχεδιαστούν τα εφαρμοστικά μέτρα, θα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Αλλά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με τη νέα νομοθεσία είναι μια πιο μέσο-μακροπρόθεσμη προσέγγιση. Τώρα, σχετικά με την κατηγοριοποίηση, την ταξινόμηση, υπάρχει και εδώ μια πρόκληση. Να τονίσω ότι στην πρότασή μας για κάποιες κατηγορίες και, και φυσικά περιλαμβάνοντας και τη νέα κατηγορία, τα on-road machinery, εκτός δρόμου μηχανήματα και οχήματα. Το λέει και η λέξη ότι είναι εκτός δρόμου, είναι σχεδιασμένα για ε, δασικές και αγροτικές εργασίες. Δεν υπόθηκε, αλλά θέλω να τονίσω ότι μετά την αλήθεια αντικτύπου για αυτή την κατηγορία αλλά και για άλλες προτείνουμε ο, ο να επιλέγει αν θέλει την έγκριση τύπου ή ε, ποια έγκριση τύπου θα επιθυμεί. Τώρα, σαν να με τα ATV, ε, η Κομισιόν έχει μια πολύ ξεκάθαρη προσέγγιση ε, Όσο οχήματα χρησιμοποιούνται για αναψυχή, κατά κύριο λόγο, ε, έχουμε μία πρόταση ε, για αυτά. Συγκεκριμένη ειδική πρόταση. Με προδιαγραφές, βασισμένα στην κατηγορία L, και η δυνατότητα να μπουν αυτά τα οχήματα στην κατηγορία T, είμαστε ανοιχτοί σε αυτό, αλλά θα πρέπει τα κριτήρια να είναι ξεκάθαρα καθορισμένα και να μην είναι έχουν στόχο να αποφύγουν τη, τη, τη, νομοθεσία. Ευχαριστώ. Αυτές είναι καλές ιδέες που θα μπορείς να λάβει υπόψη το κύριο Σπαντζέρη. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη κατηγορία. Έχουμε πέντε ομιλητές και μετά θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. έχουμε τώρα την κύριο Γκότσεν, την Γενική Γραμματεία της ΦΙΤΖΙΕΦΟ, που είναι πολλά χρόνια συμμετέχει στις επιτροπές μας. Και ο κύριος Τι ε, Το έχω το πρόγραμμα. έχουμε πει στον πρόεδρο τη της Ένωσης για τα ευρωπαϊκά αγροτικά οχήματα. Και έχουμε αντασμιλήσει για τα για τα Τέλος να αναφερθούμε και στον στο Στέφανο Μπόι, ο οποίος είναι με, μέλος στο Τμήμα Ασφαλείας και Υγείας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Συνδικάτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν που μας δώσατε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε σήμερα τη θέση μας σε σχέση με την πρόσβαση στο OBD, επισκευές συντήρηση και πληροφορίες για τους ανεξάρτητους χειριστές. Να παρουσιάσω τις δύο ομοσπονδίες. Η ΦΙΤΣΙΕΦΑ είναι η Διεθνής Ομοσπονδία των ε, Διανομέων μετά την αγορά των αυτοκινήτων. Είμαστε ανεξάρτητοι έμποροι χονδρικής λιανικής ε, για τα εξαρτήματα. Ε, και η ΕΤΖΙΑ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για Εξοπλισμούς Γκαράζ. Έχουμε κατασκευαστές, εισαγωγής διαγνωστικών εργαλείων, ε, εξοπλισμών δοκιμών και γκαράζ. Ο δόκτωρ Όλσεν αρρώστησε σοβαρά χθες, ήταν να έρθει και τον αναπληρώνω εγώ σήμερα. Η αποστολή μας από το 56 και το 80 αντίστοιχα, ο στόχος μας ήταν πάντοτε η διασφάλιση ελεύθερου και αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή ε, μεταγορά Και η Φιτζέφα και η Αιτζία συμμετείχαν στις συζητήσεις ε, για το νέο κανονισμό, για τα, την πέδηση, το Euro 5 και το Euro 6 για βαρέα οχήματα ε, πρώτη, ας πάμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Συμμετείχαμε λοιπόν πολύ στις συζητήσεις ε, επί αυτών των νομοθετημάτων και είδα εδώ πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχαν επίσης στο σχεδιασμό του κανονισμού και ακόμα εμείς ε, λειτουργούμε με τις δικές σας διατάξεις έτσι όπως τις διαμορφώσατε και είμαστε ευγνώμονες για αυτά τα νομοθετήματα. Έχουμε λοιπόν ε, εργαλεία για πολλές ε, μάρκες. Επίσης ε, έχουμε ανταλλακτικά τα οποία δίνουμε στους εξουσιοδοτημένους και τους ανεξάρτητους επισκευαστές. Πριν μπούμε στη, στην πρόσβαση στην τεχνική πληροφορία, θα παρουσιάσω την αλυσίδα της μεταγοράς, γιατί πιστεύουν καμιά φορά πολύ όταν μιλάμε για πρόσβαση τεχνική πληροφορία, μόνο για επισκευαστές, αλλά όλη η αλυσίδα περιλαμβάνει πολλούς ε, παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη συντήρηση και επισκευή των δασικών και γεωργικών οχημάτων. Δεν είναι αυτός σκοπός αυτός, αλλά για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής ε, συμμόρφωσης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος. Πρέπει να καλύπτουν ε, χαρακτηριστικά ασφάλειας και περιβαλλοντικά και όταν είναι καινούρια, αλλά και κατά τη διάρκεια όλης της ζωής που θα επισκευάζονται και θα συντηρούνται. Έχουμε κατασκευαστές διαγνωστικών εργαλείων, έχουμε χονδρέμπορους εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και εξουσιοδοτημένους ε, επισκευαστέ πολλών ε, τύπων. Δεν τα βλέπετε μέχρι κάτω στη διαφάνεια, αλλά τι χρειάζεται για τη σύγχρονη συντήρηση και επισκευή δασικών και γεωργικών οχημάτων. Υπάρχουν τέσσερα στοιχεία ή πυλώνες. Η κλασική ε, πληροφορία για τις επισκευές που περιλαμβάνει, οι πληροφορίες για το όχημα, ούτως ώστε να ταυτοποιείται αδιαμφισβήτητα, τα ανταλλακτικά και πώς θα πρέπει να τοποθετούνται σωστά, Υπάρχουν πληροφορίες για την ε, συμβατότητα OBD, χρειάζεται εκπαίδευση, κατάρτιση, χρειάζεται, χρειάζονται και εργαλεία και ε, kit δοκιμών για πολλούς τύπους οχημάτων, πολλές μάρκες και θα πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα για πλήρη λειτουργικότητα όλων αυτών των δοκιμών και συσκευών. Υπάρχουν επίσης και αποκλειστικά ε, εργαλεία που ταιριάζουν μόνο σε μια μάρκα οι ανεξάρτητοι, όμως οι επισκευαστές χρειάζονται τα πολλαπλά εργαλεία γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν τα αποκλειστικά εργαλεία από κάθε ένα χωριστά κατασκευαστή. Γιατί η πρόσβαση στην τεχνική πληροφορία είναι τόσο σημαντική, διαφοροποιείται από το Euro 5 ή Euro 6. Το σέρβις και οι διαδικασίες επισκευής για γεωργικά και δασικά οχήματα είναι ουσιαστικά τα ίδια όπως για τα εμπορικά ε, οχήματα ή επαγγελματικά και καλό τα, τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν τις αρχές αυτές γιατί μιλάμε για το κομμάτι της συναπόφασης. Πρέπει να, να ε, υποστηρίξετε λοιπόν τις αρχές για την πρόσβαση τεχνική, στην τεχνική πληροφορία όπως προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το, σε, στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματο. Επίσης πρέπει να σας πω ότι τώρα συζητάμε για τα βαρέα οχήματα, στα εφαρμοστικά μέτρα, τις λεπτομέρειες. Και όταν μιλάμε για λεπτομέρειες ε, για τα γεωργικά ή δασικά οχήματα, μπορούμε να ωφεληθούμε από το εγχείρημα αυτό το τωρινό στα εφαρμοστικά μέτρα όπου συζητάμε χαρακτηριστικά όπως προσαρμογή του ε, πελάτη ή αναπρογραμμα... Ε, αναπρογραμματισμού και μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτή τη διαδικασία στα βαρέα οχήματα ε, και στα γεωργικά και τα δασικά. Όμως, ε, και αυτή είναι η δεύτερη παύλα, η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών, των ε, πολλαπλών εργαλείων, της πληροφορίας για τη συντήρηση και τη επισκευή είναι κρίσιμη. Χρειάζονται δυνατότητες γρήγορης επισκευής για να επισκευάζονται και σε απομακρυσμένες περιοχές αυτά τα οχήματα. Εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα στο χωράφι ή στο δάσος. Εκεί θα πρέπει να έρχονται με αυτά τα πολλαπλά kit και εργαλεία για να τα επισκευάζουν όποια, όποιο τύπο η μάρκα και να έχουν. Ποιες είναι οι σημερινές τάσεις στην αγορά. Ε, μικρό η αγορά είναι εξειδικευμένη, μικρότεροι, λιγότεροι λοιπόν παράγοντες, άρα πρέπει να μπορούν να φέρνουν ε, να αντιμετωπίσουν όλες τις μάρκες. Υπάρχει αυξανόμενος αριθμός οχημάτων που είναι εξοπλισμένοι ε, με συστήματα OBD. Και τώρα προσπαθούν να ε, λάβουν υπόψη τους τα καινούρια υψηλής τεχνολογίας. Έχουν λοιπόν συστήματα OBD, συγγνώμη για την ε, ειδική αργό, δηλαδή on-board diagnostics, που σημαίνει σύνθετες επισκευές και συντήρηση και υπάρχουν και ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου ECU πολύ, πολύ υψηλής τεχνολογίας που ελέγχουν τη διαχείριση του κινητήρα, αυτόματη μετάδοση, ABS, air conditioning, πάνελ οργάνων και το, το, πανό, το, το ταμπλό κλπ. Λόγω των ε, βελτιώσεων στη τεχνολογία των οχημάτων, η κατηγορία TAF είναι, ε, ε, έχει κομπιούτερ στους τροχούς. Ναι, στο σύγχρονο όχημα τα καθήκοντα επισκευής και συντήρησης σημαίνει ότι πρέπει να διαβάζουμε λάθος κωδικούς, να τους διαγράφουμε ε, πραγματικά δεδομένα, προσαρμογές, ενεργοποίηση ε, στοιχείων, παράμετροι, ε, ρυθμίσεις παραμέτρων κλπ. Χρειάζονται λοιπόν διαγνωστικά εργαλεία πολλών τύπων. Έτσι λοιπόν η, πληρο... η πρόσβαση στην τεχνική πληροφορία και στα ανταλλακτικά είναι κρίσιμη. Ε, υπάρχει ανάγκη να στηριζόμεθα σε τυποποιημένη διαγνωστική ε, πληροφορία από το σύστημα OBD. Πρέπει να χρησιμοποιείται ε, ενημερωμένη, επικαιροποιημένη ε, διαγνωστική πολλών τύπων για να γίνεται σωστή συντήρηση και επισκευή των οχημάτων αυτών. Η πρόσβαση, πρόσβαση σε τεχνική πληροφορία ε, για όλους τους όσους λειτουργούν στον τομέα της μετααγοράς για πολλούς τύπους. Η Φιτζιέφα και η ΕτζΕα χαιρετίζουν λοιπόν τις αρχές της διατάξης όπως έχουν προδιαγραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βοηθούν να υπάρξει αποτελεσματικός ανταγωνισμός και ελεύθερη επιλογή στα προϊόντα μετά ε, την αγορά και το σέρβις καθ' όλη τη διάρκεια ε, της ζωής, του κύκλου ζωής των οχημάτων. Να αναφερθώ σε αυτό που είπαμε και πριν, εμείς είμαστε υπέρ των διατάξεων αυτών, γιατί είναι συνεπής νομοθεσία, ένα συνεπές νομοθετικό βήμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εισαγάγει παρόμοιες διατάξεις όπως έχουμε στο Euro 5, Euro 6 για τα βαρέα οχήματα κατηγορίες, ε, κατηγορίας L στα δασικά και γεωργικά οχήματα. Γιατί ε, ο κανονισμός ε, με την εξαίρεση είναι σημαντικός. Τώρα έχουμε κομπιούτερ επί τροχών εποχούμενους υπολογιστές και είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο αποκλειστικά ε, εργαλεία και δεν πρέπει να καθυστερήσουμε στην πρόσβαση στην τεχνική πληροφορία. Σας καλούμε σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν να στηρίξετε ε, απόλυτα την, την προσέγγιση αυτή όπως παρουσιάζεται στα άρθρα 47 μέχρι 49. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας πίεσα διότι ο, ο Κώστας έδωσε περίπου δύο λεπτά παραπάνω στην αρχή πριν ξεκινήσει το ρολόι, αλλά εντάξει, προσπαθήσατε, τα καταφέρατε. Επόμενος. Όλο με τα χαρτιά μου. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ρίκτερ, επόμενο. Merci de nous avoir invités à, participer à vos, à vos Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας καλέσετε να συμμετάσχουμε. Η Κλιμάρ δημιουργήθηκε το 1953, εκπροσωπεί σήμερα 17 χώρες, εντάχει 23.300 διανομής, 36.000 βάσεις σε όλη την επικράτεια που βλέπετε στη διαφάνεια και περίπου 200.000 μισθωτούς κάποια στοιχεία βασικά για να σχηματίσετε μια ιδέα όσον αφορά τις επιχειρήσεις που αντιπροσωπούμε. Η μέση επιχείρηση έχει τζίρο 4 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα αναφερθώ εκτενώς σε όλα τα σημεία του κύκλου εργασιών. Όσον αφορά τους μισθωτέους, η μέση επιχείρηση έχει 18 μισθωτούς. Το πιο σημαντικό προσωπικό μιας επιχειρήσης διανομής και επισκευών γεωργικών μηχανημάτων βρίσκεται στο εργαστήριο, στο γκαράζ με 10 μηχανικούς. Θα έλεγα ότι η επιχείρηση διανομής συνδέεται συμβασιακά με έναν κατασκευαστή, με τους πιο σημαντικούς κατασκευαστές και οι κατασκευαστές επιβάλλουν κάποιες ε, υποχρεώσεις, κυρίως και είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα μας όσον αφορά τη συνεχή κατάρτιση των μηχανικών. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και να το έχετε υπόψη σε όλη την παρουσίαση διότι είναι σχεδόν το πιο σημαντικό στοιχείο στη συζήτηση. Θέλω να μας επιστήσουμε την προσοχή στην επόμενη διαφάνεια τώρα, στις διατάξεις του κεφαλαίου 16, άρθρα, τα, στα άρθρα που αναφέρονται και αφορούν την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες στους ανεξαρτήτους επισκευαστές. Ε, διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυτές οι διατάξεις απορρέουν από τα αυτοκίνητα η ίδια διατύπωση είναι εξάλλου. Στόχος σίγουρα είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα, όμως από ό,τι γνωρίζουμε δεν υπάρχουν επισκευαστές ανεξάρτητοι που ε, επισκευάζουν πολλών εταιριών τα μηχανήματα. Έχουμε διανομής που συνδέονται συμβασιακά με έναν κατασκευαστή. Λοιπόν, αυτή η πρόταση είναι προσαρμοσμένη στον τομέα. Ε, θα θέλαμε λοιπόν να αναφέρουμε τρία σημεία όσον αφορά τις διαφορές. Όσον αφορά την ε, διάθεση της αγοράς, τεχνολογικές διαφορές και την χρήση. Δεν είναι νομική ανάλυση. Είναι οικονομικές και πρακτικές στοιχείες που αναφέρουμε εδώ όσον αφορά τις διατάξεις που ισχύουν. Λοιπόν, να πω, να σας δείξω ποια είναι η αγορά τα τρακτέρ είναι περίπου 165.000 που πολλούνται το χρόνο στην Ευρώπη και βλέπετε τα οχήματα που είναι 16 εκατομμύρια οχήματα, αυτοκίνητα που πολλούνται. Ε, η Γαλλία είναι πισωματική αγορά στην Ευρώπη, 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα για 35.000 ε, τρακτέρ. Καμία σχέση δεν έχουν οι όγκοι των πωλήσεων. Ο κύριος Ρίχτερς, ο προλαλής σας, σας είπε ότι υπάρχουν 450 είδη ε, αγροτικών αυτοκινήτων, ενός αυτοκίνητα, Ε, υπάρχουν κάποιες αναλογίες μεταξύ μικρότερου μεγαλύτερου μοντέλου. Είναι πολύ σημαντική τεχνολογία που τοποθετείται. Τα γεωργικά αυτοκίνητα, ε, οχήματα και μηχανήματα είναι υψής της τεχνολογίας ε, μηχανήματα. Άρα η συντήρηση και επισκευή ε, είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι για τα δικά οχήματα με μειωμένη αγορά. Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι τάχιστες και σημαντικές και όπως σας έλεγα πριν αυτό οδηγεί σε μια υποχρέωση κατάρτισης των μισθωτών των επιχειρήσεων, των υπαλλήλων. Οι κατασκευαστές έχουν υψηλό βαθμό απαιτήσεων στον αφορά τους διανομής τους επ' αυτού και αυτό είναι σημαντικότατο και αναφέρεται στη σύμβαση και το προσωπικό θα πρέπει να καταρτίζεται και αυτό είναι μέρημνα των επιχειρήσεων. Πέρα από την επικοινωνία και την ενημέρωση, να έχει υπαλλήλου οι οποίοι να είναι ε, ικανοί, ε, καταρτισμένοι και αρκετά περίπλοκο να το πετύχει κανείς αυτό σε όλες τις χώρες. Η αυτοδιαγνωστική είναι κάτι που αναφέρθηκε, απαιτεί μεγάλε σχετικά επενδύσει για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, όπω είναι οι επιχειρήσει που εκπροσωπώ, και διαπιστώνουμε εν γέννη ότι οι ενεξάρτητες επιχειρήσεις επισκευών μικρού μεγέθους έχουν την τάση να μειώνονται και λόγω της περιπλοκότητας του χαρακτήρα και λόγω του προσωπικού που δεν μπορούν να βρουν. Επόμενη διαφάνεια σας παρακαλώ. Προσέξτε το εξής. Χρήση του γεωργικού υλικού δεν είναι καταναλωτικά αγαθά, αντίθετα από τα αυτοκίνητα, είναι επενδυτικά αγαθά. Χρησιμεύουν ως παραγωγικές επενδύσεις των γεωργών που είναι επαγγελματίε. Μιλάμε για επιχειρήσεις γεωργικές και δασικές. Η γεωργία λοιπόν χρειάζεται, ο γεωργός χρειάζεται πάρα πολύ σημαντικές υπηρεσίες, κυρίως την περίοδο της ε, σοδιάς. Είναι πολύ απαιτητική όσον αφορά την αποτελεσματική επισκευή και τη γρήγορη επισκευή, έχει τέτοιες απαιτήσει. Ε, απ' την άλλη όσον αφορά τη γεωγραφική πτυχή και τη ανομή των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις βρίσκονται στην Ήπεθρο, δεν υπάρχει γεωγραφική συγκέντρωση, αλλά χρειάζεται ένα δίκτυο εδαφικό πολύ σημαντικό για να εξασφαλίζεται ποιοτική παροχή υπηρεσιών και τέλος να διευκρινίσω ότι το αγροτικό υλικό είναι οχήματα που πηγαίνουν στο δρόμο αλλά έχουν χρήση στη δουλειά και είναι ενδεχομένως επικίνδυνα μηχανήματα. Δηλαδή κάθε χρόνο ε, ε, έχουμε ατυχήματα στη, λόγω της χρήσης αυτών. Λοιπόν, είναι, χρειάζεται και ενημέρωση αλλά έχουμε, που μπορεί να δοθεί στους πάντες, αλλά έχουμε πρόβλημα στον αφορά τις επισκευές και τη συντήρηση, όπως σας είπα. Λοιπόν, εν κατακλείδη, οι διατάξεις του κεφαλαίου 16 α, δεν θα έχουν θετικές συνέπειες για τους πελάτες μας, τους αγρότες. Ο αγρότης κινδυνεύει να έχει μια υπηρεσία συντήρησης και επισκευής ε, ε, ε κατωτέρου επίπεδου. Αυτές οι διατάξεις για τη διαβίωση των πληροφοριών είναι επικίνδυνο, επικίνδυνο τον τελικό χρήστη και είναι πολύ ε, δαπανηρά μέτρα αυτά που επιβάλλονται μέσω των διατάξεων για τις επιχειρήσεις αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Τα μέλη σας είναι ανεξάρτητοι επισκευαστές. Και εκείνοι που έχουν franchise, έτσι. Ναι, ναι, είναι η απάντηση. Ναι, ναι, δίκιο έχετε. Αυτό είναι. Ουσιαστικά είναι, έχουν franchise. Εχωρούνται δικαιώματα ανεξάρτητες επιχειρήσεις και λοιπόν έχουν αυτό, αναλαμβάνουν, τους αναθέτει η κατασκευάστη εταιρεία. Τις επισκευές έχουν franchise. Τα μέλη σας είναι εγκεκριμένοι επισκευαστές για κάποιο κατασκευαστή. Θα μπορούν να επισκευάζουν πολλές μάρκες, αλλά έχουν franchise από τον κατασκευαστή. Απάντηση. Είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις που δένονται με έναν κατασκευαστή. Οι περισσότερες και επειδή υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία προϊόντων, η επιχείρηση που διανέμει το αγροτικό υλικό έχει υποχρέωση να προτείνει, για να προτείνει την καλύτερη υπηρεσία και το καλύτερο προϊόν για τον πελάτη να έχει πολλούς κατασκευαστές, αλλά όχι στο ίδια γκάμα προϊόντων. Μπορεί να έχει έναν κατασκευαστή τρακτέρ, άλλο κατασκευαστή που σου δίνει αυτόν που δημιουργεί κονιορτοπή, ε, καταστροφέα μάλλον, ε, Οπότε υπάρχει σύμβαση με τον κατασκευαστή για κάθε είδους ε, μηχάνημα, για διαφορετική χρήση. Ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο κύριος Τζένκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Δεν θα περάσω όλες τις διαφάνειες, γιατί οι περισσότερες είναι για θέματα που έχουν καλυφθεί ήδη τους προλαλισσάντες θα ε, σας πω για τις δύο πρώτες διαφάνειες. Θα μιλήσω ελεύθερα. Έχω την αίσθηση σήμερα ότι υπάρχει λίγο σύγχυση μεταξύ ε, των, αυτοκινήτων και, των, ε, και της βιομηχανίας και οχήματα. Ένα τρακτέρ δεν είναι αυτοκίνητο. Βέβαια έχει τέσσερα αυτοκίνητα, ε, συγγνώμη τέσσερις τροχούς, αλλά όπως βλέπετε, το τρακτέρ είναι ένα πολυτουργικό όχημα που έχει διάφορα εξαρτήματα. Μπορείτε να δείτε στη διαφάνεια. Και είναι πλέον ένα εργαλείο για τους αγρότες, με το οποίο ζουν οι αγρότες από αυτό. Αν χαλάσει το τρακτέρ, δεν μπορείς να βγάζεις άλλα λεφτά. Ενώ αν χαλάσει το αυτοκίνητό σου, μπορείς να πάρει το λεωφορείο. Να υπογραμμίσω αυτό. Οι πελάτες είναι πολύ απαιτητική. Ε, δεν είναι τόσο καλοί πελάτε όμως γιατί το εισόδημά του είναι πολύ μικρό σχέση με το μέσο εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε σαν διαφορά με την βιομηχανία αυτοκινήτων. Ε, προτινόμενος κανονισμός βασίζεται στην υπόθεση ότι είμαστε ένα κλάδο τη ε, αυτοκινητικής, βιομηχανία που δεν είμαστε. Να σας δώσω τώρα κάποιους λόγους, γιατί ζητάμε το Κοινοβούλιο να απαλείψει το κεφάλαιο 16 και, το, και τα άρθρα 47-50. Επιπλέον, σαν κατασκευαστές, ε, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι ανεξάρτητοι επισκευαστές οι οποίοι λειτουργούν. Θα ήθελα να δούμε βέβαια τα νούμερα που υπάρχουν. Τώρα η οργάνωσή μας, η ΣΕΜΑ, έχει πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα για το κεφάλαιο 16. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχει γίνει μια μελέτη αντικτύπου. Δεν μπορούσαμε ξαφνικά να αλλάξουμε το σύστημα διανομής από τη μια μέρα στην άλλη, χωρίς να έχουμε μια μελέτη αυτό. Δεν μπορούσαμε να αξιολογεί την δυναμική της αγοράς. Πρώτον αυτό. Δεν, είχαμε, δεν μπορούσαμε να εκφραστούμε πάνω σε αυτό και δεν γνωρίζαμε ότι είχε γίνει κάποια μελέτη αντεκτύπου και αν είχε γίνει πάνω στο κεφάλαιο 16 του κανονισμού. Ε, μπορεί να έχει γίνει. Πάντως δεν είχε λάβει υπόψη τις ανάγκες της βιομηχανίας και θεωρούμε ότι α, όλο αυτό αντιβαίνει στα, στα, συμφέροντά μας. Επιπλέον θεωρούμε ότι η πρόταση βασίζεται σε μια λα, λανθασμένη νομική βάση γιατί βασίζεται στο άρθρο 114 το τρακτέρ πάντα ε, ήταν διαχωρισμένο από, την, από το αυτοκίνητο και ποτέ δεν είχαμε τον ίδιο νομική βάση. Ε, στην νομική βάση στο 330 που αναφέρθηκε, 340, υπάρχουν τεράστιες διαφορές γιατί στα αυτοκίνητα υπάρχουν επιλεκτικοί dealer, ενώ εμείς έχουμε ε, αποκλειστικούς dealer. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει τη μία μέρα στην άλλη. Εδώ και 40 χρόνια υπάρχει αυτό το καθεστώς, δεν μπορεί να αλλάξει έτσι ξαφνικά. Και θα θέλαμε ε, οποιασδήποτε μελλοντικέ διατάξεις που θα βασίζονται στο άρθρο 114 της συνθήκης, η οποία είναι ξεκάθαρη, Έχουμε λοιπόν εδώ ένα άρθρο, το 101 και το 102 της συνθήκης, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται στο άρθρο 103 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι σημαντικό ότι δεν είμαστε στο ίδιο νομικό πλαίσιο, να το τονίσουμε αυτό. Ε, επίσης υπάρχει η δομή των αυτό που θα λέγαμε στα γαλλικά, η οικονομία του συμβολέου. Υπάρχει αυτή η δομή του, της αγοράς σε αυτό το θέμα. Αν μας, ε, ο νόμος μας, ε, μας επιβάλλει να δώσουμε αμέσω πρόσβαση στα OBD, τότε θα είμαστε αντίθετοι με τα συμβατικές μας υποχρεώσεις. Μια άλλη νομικό πρόβλημα είναι το, το κεφάλαιο 16, το οποίο δημιουργεί ε, μια επιπλέον υποχρέωση που οδηγεί σε μια διπλή ε, διαδικασία για τα πρόστιμα. Μπορεί να πάρεις να, δύο φορές πρόστιμο για, το ίδιο, για την διαπαράβαση. Το ένα σύμφωνα με το κεφάλαιο 16, το οποίο θέτει νέες κυρώσεις για τους κατασκευαστές που δεν παρέχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά επιπλέον θα μπορούσες να πάρεις ένα πρόστιμο σύμφωνα με, το, με τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ε, είναι άδικο. Και τελικά αυτά τα πέντε σημεία, η έλλειψη με της τύπου, η λάθος νομική βάση, η δομή και το θέμα της ε, θεματικής υποχρέωσης, και το κεφάλαιο 16 το οποίο δημιουργεί ε, ένα, μια υπερκάλυψη. Αλλά επιπλέον σε οικονομικό επίπεδο θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση για τους πελάτες, καμία εγγύηση ότι θα παρέχονται καλύτερες υπηρεσίες. Αντιθέτως θεωρούμε ότι με τις ανεξάρτητους επισκευαστές μπορεί να κάνουν ε, ε, ε, επιλεκτική δουλειά, να επικεντρωθούν στα πιο ωφέλιμα σε αυτούς σημεία, και, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένας επισκευαστής πρέπει να παρέχει όλες τις, τις επισκευές, είτε είναι ε, συμφέρουσες είτε όχι, και να είναι και 24 ώρες βάση. Όταν ε, τα μεσάνυχτα ξαφνικά χαλάσει το τρακτέρ σου, δεν θα βρεις κάποιον να σου επισκευάσει το όχημα του, που είναι ζωτική σημασία για πολλούς αγρότες. Τα ανταλλακτικά αυτά επίσης θα ε, εισάγονται τα περισσότερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση, οπότε δεν θα υπάρξει και κάποια ωφέλο για την αγορά. Δεν θα υπάρξει επίσης για τον dealer, ε, για τον αντιπρόσωπο όφελος. Ε, σε σχέση με, την Ευρωπαϊκή, με τις ΗΠΑ και τον Καναδά έχουμε πολύ περισσότερους αντιπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το κεφάλαιο 16 θα, θα αυξήσει την τάση μείωση των αντιπροσώπων και θα οδηγήσει σε λιγότερε υπηρεσίε παρεχόμενε, αλλά και λιγότερη απασχόληση στον κλάδο. Δεν θα υπάρχει κανένα όφελος επίσης για το, για το περιβάλλον. Ε, θα δοθεί ευκαιρία να, να μην ε, υπάρχει σωστός έλεγχος στα θέματα των εκπομπών, της ασφάλειας. Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι το κεφάλαιο 16 θα διαταράξει το, την αγορά, δεν θα βοηθήσει σε θέματα ασφάλειας. Και γι' αυτό η ΣΥΜΑ ζητάει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να το, το κεφάλαιο 16 και σας ζητούμε να βρείτε κάποιον άλλον τρόπο να νομοθετήσετε ε, και να, ε, να και δημιουργήσει δημιουργήσετε το κανονιστικό πλαίσιο για αυτά τα, για αυτά τα οχήματα. Ευχαριστώ. Uh, Θα δοθεί ευκαιρία αργότερα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Μάρης για να δούμε εάν θα ασχοληθεί και εκείνος με το θέμα αυτό και αν συμφωνεί με τον προηγούμενο μιλητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είμαι θα πολύ ευτυχής ως ε, καταναλωτές που ε, για το γεγονός ότι προσκληθήκαμε εδώ. Η ΣΕΤΑΡ είναι η ε, συμμετοχή εργολάβη στον τομέα αυτό, γιατί δεχόμαστε εργολαβίες, αναλαμβάνουμε εργολαβίες στον τομέα και εκπροσωπούμε περίπου 100.000 επιχειρήσεις. και καλύπτουμε 500.000 ε, πρόσωπα. Η συμβολή μας είναι σημαντική για τους γεωργούς και ο ετήσιος τζίρος μας ε, είναι περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ο κύκλος εργασιών αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο χάρη στην μεγάλη χρήση πολλές φορές μεγάλων μηχανημάτων. Εδώ μπορέσαμε λοιπόν να δώσουμε μια μεγάλη συμβολή ε, στις εκμεταλλεύσεις αυτές. Αυξήσαμε δηλαδή την ανταγωνιστικότητα. Οι ετήσιες επενδύσεις είναι σημαντικές. 8 δις ευρώ επενδύονται για νέα μηχανήματα. Θεωρούμε ότι είμαστε η σημαντικότερη ομάδα χρηστών των δρόμων. Δραστηριοποιούμεθα επίσης και στην γεωργία, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πολλές φορές πρέπει να μεταφέρουμε οδικά τα μηχανήματα αυτά και μας ενδιαφέρει υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Να προσθέσουμε ότι τις προηγούμενες ε, δεκαετίες οι διασυνοριακές μεταφορές αυξήθηκαν πολύ και γι' αυτό ε, συμβάλαμε και εμείς. Είναι πολύ σημαντική η ε, εξειδίκευση των γεωργικών μηχανημάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι τα μηχανήματα αυτά δεν ε, πρέπει να ε, αντιστοιχούν στις εθνικά συστήματα έγκρισης τύπου, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και να καλύπτουν τους όρους και προϋποθέσεις που θέτουν και άλλες χώρες. Το τα σημαντικότερα στοιχεία αναφέρονται στον κανονισμό, εναρμόνιση της παραγωγής, των γεωργικών μηχανημάτων, των ελκυστήρων, Επίσης θέλουμε ενιαίους κανόνες ώστε τα μηχανήματα αυτά να ε, κυκλοφορούν στους δρόμους με μεγαλύτερη ασφάλεια και θέλουμε με απλούστερες νομικές διατάξεις να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Η ασφάλεια. Η ασφάλεια συνδέεται με καλά συστήματα πέδησης. Πρέπει επίσης να αναφέρομαι στο σχέδιο κανονισμού την συμβατότητα μεταξύ των μηχανημάτων και των ελκυστήρων ε, είναι σημαντικό αυτό. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότερη παραγωγή των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιούνται με αποδοτικότερο τρόπο και στο χωράφι, και στο, και στο χωράφι και στο δρόμο. Με βάση τον κανονισμό πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής. θα πρέπει να είναι απλούστερη διαδικασία έγκρισης όχι μόνο για τα ε, καινούρια αλλά και τα μεταχειρισμένα μηχανήματα γιατί όλα και, όλο και περισσότερα χρησιμοποιούνται διασυνοριακά και μετά ε, χρησιμοποιούνται σε άλλη χώρα ως μεταχειρισμένα και για τα ρημουλκούμενα χρειάζονται νέοι κανόνες και για τα, ε, ε, ε, το ρημουλκούμενο εξοπλισμό. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για ε, μια ασφαλέστερη χρήση και στο δρόμο και αλλού συχνά λέμε ότι υπάρχουν εξοπλισμοί που δεν ε, πληρούν τις ε, προδιαγραφές κάποιων κρατών μελών. Επίσης, ε, αναφέρει ο κανονισμός και το είπαν και άλλοι ομιλητές, τα, τον κινητό εξοπλισμό, τα κινητά μηχανήματα αυτά τα κινητά μηχανήματα παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μηχανήματα με πολύ εξειδικευμένους τομείς εφαρμογής που αυξάνουν όμως την ανταγωνιστικότητα αυτά τα, αυτή η κατηγορία ειδικών μηχανημάτων θα πρέπει να αναφερθούν ε, ιδιαίτερα στον κανονισμό. Επίσης, ε, πρέπει να πω ότι και στο τομέα των οικοδομών χρησιμοποιούνται, έχουν δηλαδή μεικτή χρήση. Μπορεί να σας εκπλήξει αυτό ε, λίγο αλλά πρόκειται για μηχανήματα διπλής χρήσεως συχνά. Με άλλα λόγια, μιλάμε για μηχανήματα σε χωματουργικά έργα, σε εγκυοβελτιωτικά έργα, ε, πολλών γεωργικών χρήσεων. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή σας σε αυτή τους την ε, ιδιότητα ως αγροτικές ε, εκμεταλλεύσεις, ε, ε, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ενδιαφέρονται για τρακτέρ ταχύτητα 40 χιλιόμετρων. Δεν θέλουμε η μεγαλύτερη ταχύτητα γιατί τα τρακτέρ δεν εκτελούν μεγάλες μεταφορές Γενικά η πρόταση είναι θετική και με κάποιες απλουστεύσεις μπορούμε να μιλήσουμε για δύο κατηγορίες, η Α και η Β με βάση την ταχύτητα και το όριο, δηλαδή κάτω και πάνω από τα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε εμείς με την πρόταση αυτή δηλαδή. Το κεφάλαιο 16 τώρα που έχει επικριθεί αρκετά. Εμείς το βλέπουμε πρακτικά το θέμα. Θέλουμε να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες και για τους χρήστες αλλά και για τους ειδικού εξειδικευμένους επισκευαστές. Αυτό είναι σημαντικό για να βελτιστοποιήσουμε κόστος επισκευών, ε, και λειτουργίας των μηχανημάτων. Στον κανονισμό και στην ιδεολογική έκθεση η Κομισιόν ε, θα κάνει κάποιες ε, τεχνικές παρατηρήσεις και διευκρινήσεις. Δεν μπορώ να κρίνω ε, τώρα το 2014 εάν είναι μία σωστή προθεσμία. Ο κλάδος, η βιομηχανία θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες προϋποθέσεις θα ισχύουν ε, για τα μηχανήματα που κατασκευάζονται θα πρέπει να συμπεριληφθούν και κινητά μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και στον τομέα των οικοδομών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρισε Τελευταίος ομιλητής, πολύ σημαντικός, ο Στέφανο Μπόι ε, από το ε, Ινστιτούτο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Chairman Arbour, uh, Rapporteur Panseri, thank you for giving Ευχαριστώ κύριε Σιγητά που, και κύριε Πρόεδρε που μας δίνει τη δυνατότητα σε συνδικάτα συμμετάσχουμε στην ε, συζήτηση. Είναι πολυνόμιο να απευθυνόμεθα σε τέτοιο κροατήριο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προλαλήσαντες για τις εντυπωσιακέ ε, πτυχές που ξετύλιξαν. Εγώ θα αναφερθώ στο θέμα ε, υγιεινής και ασφάλειας. Υγιεινής και ασφάλειας. Τα σχόλιά μου και η παρουσίασή μου έχουν σαν σχόλιο να μοιραστώ μαζί σας σκέψεις για την υγεία και ασφάλεια. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι σχετικά με αυτό συγχαίρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά που έκανε και πιο συγκεκριμένα τον επικεφαλή της μονάδας, ε, της αρμοδίας, το προσωπικό του, της μονάδας για τα οχήματα και τα αυτοκινήτα. Πιστεύουμε ότι η πρόταση είναι ένα έξοχο έγγραφο για τη διάσταση αυτή της υγείας και της ασφάλειας ε, καλωσορίζουμε τη ρητή αναφορά της ασφάλειας στον τόπο εργασίας, βασικό στοιχείο της προτάσεως. Έχω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες συστάσεις πώς θα μπορούσε να εμπλουτιστεί εν λόγω πρότασης για την επίτευξη των στόχων. Το άρθρο 8 δείχνει θεμελιώδεις πτυχές της υγιεινής και ασφαλείας που θα πρέπει τις προϋποθέσεις αυτές, προδιαγραφές να τις εφαρμόζουν οι κατασκευαστές ε, πτυχέ που καλύπτονται από διάφορε οδηγίε. Πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Αν θέλουμε να πετύχουμε του στόχου τη προτάσεω, θα πρέπει να έχουμε μια σειρά απαραίτητε πτυχέ. Οποιοδήποτε μηχάνημα που χρησιμοποιείται στον τόπο εργασία θα πρέπει να καλύπτονται αυτέ τι πτυχέ. Βλέπετε, για τη βιομηχανία τίποτα δεν είναι καινούριο. Ήδη οι πτυχέ λαμβάνονται υπόψη από αυτού που θέλουν να συμμορφωθούν, από τι επιχειρήσει που θέλουν να συμμορφωθούν αλλά το να αναφέρονται ρητά στην πρόταση θα μπορούσε να βοηθήσει ε, ότι θα επικρατούν ισότιμε συνθήκες για το τομέα. Γιατί? Γιατί οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν μπορούν να διακινδυνεύσουν ανταγωνισμό ει βάρος ασφαλείας. Είναι λογικός ανταγωνισμός και αναγκαίο. Αλλά όχι σαν τίμημα να έχουμε την ασφάλεια. Στα χρονικά όρια που έχω στη διάθεσή μου δεν μπορώ να τεκμηριώσω, να υποστηρίξω Κάθε γραμμή που παρουσιάζω, κάθε πτυχή ασφαλείας όμως, προτιμώ να δώσω λεπτομέρειες επί μίας από αυτές. Το ROPS, το Rollover Protection Systems, δηλαδή τα συστήματα που ε, προστατεύουν σε περίπτωση ε, που του μπάρει το όχημα. Ε, ελαχιστοποιούνται έτσι ε, τα, οι συνέπειες του αν του μπάρει το τρακτέρ. Τα τρακτέρ όμως χρησιμοποιούνται πολύ συχνά σε περιπτώσεις όπου ε, δεν θα, θα εμπόδιζε ένα τέτοιο μέτρο για την προστασία για τις τούμπες στη δουλειά και υπάρχουν αποσυρώμενα συστήματα τέτοια προστασίας. Θα πρέπει να διπλώνονται αυτά όμως τα συστήματα από τη στιγμή που έχει τελειώσει η χρήση. Όποτε χρειάζεται θα μπορούν να ανεβαίνουν αυτά τα συστήματα προστασίας όταν μπαίνουμε και περνάμε από κάποιο, κάτω από κάποιο εμπόδιο. Πολύ συχνά ε, σε μοιραία ατυχήματα έχουμε ανατροπή του, ε, του ε, ελκυστήρα και έχουν μείνει μαζεμένα τα συστήματα και κλειδώματα προστασίας, ο κλωβός προστασίας. Γιατί είναι πολύ συχνά δύσκολο να κάνει κανείς ελιγμούς με αυτά. Γιατί. Ρωτήστε τον εργαζόμενο και θα σου εξηγήσει. Θα σου λέει αν πρέπει συχνά να ανεβάζω και να κατεβάζω, είναι δύσκολο να δουλέψω. Η απάντηση είναι ότι είμαστε επαγγελματίε, είμαστε λογικοί, ε, αλλά είμαστε επίσης ε, αντικείμενα λαθασμενη χρήση αυτών των μέσων. Ήδη υπάρχουν λύσεις στην αιχμή τη τεχνολογία. Είναι προβλέψιμη η λανθασμένη χρήση. Γιατί το λέμε αυτό. Ρωτήστε τον εργαζόμενο. Μπορούμε να το προβλέψουμε. Εγώ δεν μπορώ, λέει ο εργαζόμενο. Δεν θέλω να το κάνω. Θέλω κάτι το οποίο να είναι γενό ασφαλέ. Και η βιομηχανία ήδη ε, διάφορε λύσει αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα λύσης, Πρόεδρε. Και αυτό το παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα σωστής εφαρμογής του άρθρου 114 της συνθήκης. Πάρτε τεχνολογική καινοτομία, εφαρμόστε την για να είναι ασφαλή τα μηχανήματα αυτά. Επόμενο, άρθρο 8 Λοιπόν, λεπτομερείς απαιτήσει της κατεξουσιοδότηση πράξης. Στον τόπο εργασίας, άμα εκφράζονται απόψεις, οι πληροφορίες που βοηθήσουν τη βιομηχανία να βελτιώσει το σχεδιασμό των ελκυστήρων. Θα πρέπει η πρόταση να συμπεριλαμβάνει αυτή τη ε, διάσταση. Αυτό είναι ένα κείμενο που υπάρχει και το προτείνουμε. Αυτή η φράση ταιριάζει σχεδόν φυσιολογικά στο κείμενο και του δίνει μεγαλύτερη ουσία. Δίνει μεγαλύτερη ουσία στον στόχο που προσπαθεί να πετύχει η παράγραφος. προσπαθώ να συνοψίσω τώρα σε διάφορα σημεία, σε διάφορους παραγράφους ανησυχίε μας. Αυτή η πρόταση μπορεί να μειώσει το κόστος των ατυχημάτων. Όχι μόνο σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και το οικονομικό κόστος ε, των ατυχημάτων στον τόπο εργασίας. Στη δεύτερη παράγραφο λέμε ότι στην κατακαιρματισμένη κοινότητα των χρηστών ελκυστήρων και αγροτικών μηχανημάτων που είναι βασικά κατακαιρματισμένη κοινότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα μπορούσαμε να είμαστε υπεύθυνοι και να βελτιώσουμε την ασφάλεια για εκατομμύρια ε, εργαζομένου. Πώ να το κάνουμε. Στη τρίτη παράγραφο λέει ότι ο φθηνότερο τρόπο για να το πετύχουμε αυτό, να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα προβλήματα, ή να τα λάβουμε υπόψη κατά τη φάση του σχεδιασμού. Ούτω ώστε να δούμε ε, τι γίνεται ε, στη, στην χρήση του μηχανήματος. του χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος το μηχάνημα. Χρειαζόμαστε πληροφορίε συνεπώ από τους εργαζόμενους. Μετά στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε διάφορες συστάσεις. Σημείο Α. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την τεχνολογική καινοτομία και να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας γεωργικών μηχανημάτων στην ε, Ευρώπη. Το σημείο Α μπορούσε να ενισχυθεί αν οι τεχνικές διατάξεις αντικατοπτρίζουν την πραγματική πρακτική, την καθημερινή δουλειά. Και το σημείο C λατινικό, εκεί η πρόταση μπορεί να βοηθήσει να κινηθούν καλύτερα τους συμμορφούμενους οικονομικούς φορείς έναντι αθέμη του ανταγωνισμού που αγνοούν ή υπερκεράζουν τους ε, ε, τους κανόνες του παιχνιδιού. Και η υποπτία της αγοράς, το σημείο C, είναι επίσης το εργαλείο που μπορεί να ε, οδηγήσει σε πιο ε, ισότιμους ελέγχους στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ίσες, οι ίδιες δράσεις εναντίον εκείνων που δεν συμμορφώνονται. Τέλος, η, η οργάνωσή μου δεν είναι μόνη της. Δημιουργούμε για να ανταποκριθούμε στο αίτημα του Προέδρου και του Συγητού να λαμβάνεται υπόψη η ανησυχία του χρήστου, δημιουργούμε δίκτυο ε, μηχανικών που προέρχεται και τις τάξεις των αρχών και των γεωργών. Να σας πω ότι εσείς, Πρόεδρε, ο εισηγητής σας, μπορείτε να βασιστείτε στο ΕΤΟΥΙ για τη διάδοση της γνώσης και ε, θα σας διαθέσουμε αυτές τις γνώσεις για να μπορέσετε να πετύχετε τους στόχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, κύριε Μπόι, για τις πολύ πρακτικές προτάσεις σας, λογικές προτάσεις σας και που ε, διαθέτεται πόρους ε, που μπορεί να χρησιμοποιήσει και ο εισηγητής και εμείς. Πριν μιλήσει ο κ. Ματίνο, κύριε Ρούλε ή ο κ. Σβάμπ, άμα θέλουν να θέσουν κάποιες ερωτήσεις εμπειρογνώμονες. Έχω και εγώ μία-δύο ερωτήσεις. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ο κ. Σβάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ομιλητές με τις εξαιρετικές ομιλίες τους, πολύ διαφωτιστικές για μας. Εγώ κατάλαβα ότι η κατάσταση στην αγορά υπάρχουν διαφορές γιατί λόγω μεγέθους αγοράς και λόγω προδιαγραφών ασφαλείας των ε, μέρων. Βέβαια δεν ξέρω αν η διαφορά μεγέθους δικαιολογεί την ύπαρξη διαφορετικών κανόνων και εις ό,τι αφορά τα στοιχεία ασφαλείας, κινητήρες κλπ. Πάλι δεν ξέρω αν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές. Ίσως ε, μπορεί να μου εξηγήσουν οι ομιλητές γιατί δηλαδή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι δύο κατηγορίες οχημάτων από τον κανονισμό με διαφορετικό τρόπο ή από διαφορετικούς κανονισμούς. Και εγώ και ο κύριος Παντσέρη, ε, βέβαια ο κύριος Παντσέρη μπορεί να ρωτήσει ό,τι θέλει όποτε θέλει να δούμε κάποια επιχειρήματα σε σχέση με τις τεχνικές πληροφορίες και την πρόσβαση σε αυτές. Υπάρχουν και ε, ε, αντιστοιχίε με τον κανονισμό για τα δίτροχα οχήματα. Αναφέρθηκε και από την κυρία Γκότσεν ότι κατηγορία ΤΑΦ γίνονται υπολογιστές εποχούμενοι και ο κύριος Τριανκούρη είπε για τα επαγγελματικά οχήματα ότι είναι απαραίτητο να είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι οι χρήστες και εκείνοι που θα έχουν πρόσβαση στην τεχνική αυτή πληροφόρηση. Ο κύριος Μάρης ε, κράτησε πιο ουδέτερη στάση, υποθέτω ότι συμφωνεί και εκείνος ότι τα μέλη θέλουν πρόσβαση η ερώτηση λοιπόν και προς τους τρεις είναι πιστεύετε ότι δεδομένου της πολυπλοκότητας των ε, εξοπλισμών αλλά και ο κυρίος Πόη ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα της ασφάλειας των μηχανημάτων και είπε σημαντικά πράγματα σχετικά με τις ε, ε, αθέλητες κινήσεις, τις λάθος κινήσεις ή την κακή χρήση των μηχανημάτων. Πιστεύετε λοιπόν ότι για να διασφαλιστεί ότι η πληροφορία θα δίδεται μόνο σε αυτούς που ασφαλούς, ασφαλώς θα την χρησιμοποιήσουν, που θα είναι καταρτισμένοι δηλαδή για να δεχτούν την πληροφορία, αυτό απαιτεί να είναι μέρος ενός εξουσιοδοτημένου δικτύου των κατασκευαστών που ήταν μια πρόταση ή είναι εφικτό και δυνατόν ο κατασκευαστής να είναι βέβαιος ότι η πληροφορία θα πηγαίνει σε ειδικού επισκευαστές που δεν θα είναι μέλος, μέλη του δικτύου, για παράδειγμα. Η δεύτερη ερώτηση αφορά στην πρόσβαση στο δίκτυο των επισκευαστών, γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτό που είπε ο κύριος ε, Ρίπτερ, είναι ότι είναι οργανωμένοι με, διαφορετική, με διαφορετικό τρόπο η διανομής ε, ε, τρακτέρ από των αυτοκινήτων ή των ε, ε, μοτοσύκλετων ή διτρόχων. Τώρα, η απάντηση που έδωσαν οι επισκευαστές διτρόχων είναι ότι πολλοί δεν θέλουν να είναι στο δίκτυο των επισκευαστών αυτοκινήτων. Αυτό είναι σοβαρό θέμα για τα τρακτέρ και ρώτησε τον κύριο Τρίγκο εάν ε, μπορώ, ε, εάν είμαι επισκευαστής εξοδοτημένος να συμμετέχω στο δίκτυο, δηλαδή επηρεάζεται ο ανταγωνισμός ε, και παίζει αυτό ρόλο στο αν θα γίνει κάποιος δεκτός στην οργάνωση ή στο δίκτυο, είναι αρκετά σημαντικό το ερώτημα. Και ο κύριος Ρίκτερ ε, είναι σημαντικό να απαντήσει και στην ερώτηση του κυρίου Σβάμπ που θα απαντήσουν και άλλοι. Ίσως ο κύριος Μπόι μπορεί να αρχίσει και μετά η κυρία Γκότσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομο σχόλιο. Έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό θέμα η χρήση της πληροφορίας και για, η διαδικασία του σχεδιασμού περιλαμβάνει και ένα πακέτο πληροφορίας που είναι κομμάτι του μηχανήματος. Βέβαια οι συνάδελφοι είναι πιο ενδεδειγμένοι για να απαντήσουν, αλλά εγώ θέλω να αναφερθώ ότι για μένα αυτό είναι ένα θέμα ασφάλειας, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας το προφίλ του τελικού χρήστη του τρακτέρ, Έχουμε μια κατακαιρμανισμένη κοινότητα όπου είτε πραγματογνωμοσύνη δεν είναι ίδια. Έχουμε ε, γεωργούς, οικογένειες, μικρές εκμεταλλεύσεις που έχουν περιορισμένη χρήση στην πληροφορία. Πρέπει να το δούμε δηλαδή αυτό το θέμα της πρόσβασης. Περιορίζομαι σε αυτό και οι ε, συνάδελφοι θα επισέλθουν σε περισσότερες λεπτομέρειες. Να τονίσω, Πρόεδρε, και πάλι, ότι δεν είμαστε τέτεροι σε αυτό. Είναι καλό η... Θα πρέπει να είναι προσβάσιμες οι πληροφορίες για την επισκευή και τη συντήρηση. Ε, οι ανησυχίε της διαφόρων μιλτών όπως τη ΣΕΜΑ δεν είναι κατανοητές σε εμάς. Είναι πολύ εξειδικευμένα μηχανήματα για τα οποία χρειάζεται τεχνογνωσία, αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι η αγορά μπορεί να λειτουργήσει εδώ. Γιατί, γιατί η, η αγορά ξεχωρίζει τα καλά μηχανήματα από τα κακά. Δεν νομίζω ότι είναι... Ε, ότι τα, μια κακή μηχανή ή ένας κακός επισκευαστής θα, έχει, θα είναι μακρόβια. Οπότε νομίζω ότι η ενας κακος επισκευαστης θα θα ειναι μακροβια οποτε νομιζω οτι η αγορα θα το χειριστεί. Λοιπόν, μην είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Να υπογραμμίσω ότι κάτι που δεν συζητήσαμε ήταν τα, πνευματικά δικαιώματα και το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει το δικαίωμα να, το, να μην ε, ε, γίνουν δημοσία τα, ε, τα εγχειρίδια επισκευής αν δεν το θέλουν. Το θέμα τώρα είναι η έγκριση τύπου, η ασφάλεια ή ο ανταγωνισμός. Αν είναι θέμα ανταγωνισμού, τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί το δίκαιο ανταγωνισμό. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό, γιατί το θέμα της πρόσβασης σε OBD έχει πρώτα καθορίστηκε από το δίκαιο ανταγωνισμό, αλλά μετά ε, περιλήφθηκε στην πρόταση έγκριση τύπου. Αν όμω μιλάμε για υγιεινή και ασφάλεια, τότε η βιομηχανία καλωσορίζει κάθε διάταξη και δεν μπορώ να μιλήσω για τη δική μα ε, εταιρεία. Έχουμε μια μακρά παράδοση ε, στο να προστατεύσουμε τα θέματα ασφάλειας, να ανταλάβουμε υπόψη μα τα θέματα ασφαλείας. Δεν είναι το θέμα ανταγωνισμού εδώ. Υπάρχουν δύο διαφορές που θα πρέπει να, να δούμε. Άκουσα επίσης, υπάρχει αίσθηση ότι τα τακτέρ δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Εγώ δεν έχω τα νούμερα, αλλά πέρσι ήμουν μια, σε ένα συνέδριο για την ασφάλεια στα τακτέρ ο αριθμός των θανάσιμων ε, ατυχημάτων είναι κάτω από 100 το χρόνο, ενώ όταν μιλάμε για αυτοκίνητα μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ε, θανάσιμα ατυχήματα. Τώρα, οπότε, είναι αστείο η, η αυτοκινητιστική βιομηχανία να μας λέει σε εμά ότι πρέπει να βελτιώσουμε τα προτεγραφές ασφαλείας. Το τρακτέρ είναι πιο ασφαλές, ασφαλώς μπορούμε να ε, να βελτιωθούμε. Αλλά ας διαχωρίσουμε τις δύο διαστάσεις. Μιλάμε για ασφάλεια ή για ανταγωνισμό. Για την ασφάλεια δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ε, υποστηρίζουμε πλήρως αυτή την πρόταση. Μπορούν να υπάρξουν βελτιώσεις στο γενικό επίπεδο. Αλλά δεν συμφωνώ, όπως ε, προείπα, στο θέμα των ανεξάρτητων ε, επισκευαστών. Τι να πω. Πολλά ζητήματα έχουν ε, ανακατευθεί στο διάλογο και θα ήθελα να βάλω μια τάξη σε διάφορα θέματα. Είπατε ότι είστε τόσο διαφορετικοί από τον αυτοκινητιστικό η βιομηχανία, αλλά έχετε προσπαθήσει να αντιγράψετε πολλά επιχειρήματα τα οποία εμεί ε, είχαμε στο Euro 5 και Euro 6 και τα επιχειρήματα που είδαμε στο διάλογο για τα επιβατικά οχήματα και τα βαρέα οχήματα. Επομένω, ας μην ανακατεύουμε τον δίκαιο ανταγωνισμό, το θέμα επιλητικής διανομής, την ε, πρόσβαση σε εξειδικευμένε ε, πληροφορίε και σε θέματα ασφαλεία. Σα μην τα ανακατεύουμε όλα. Το σύστημα επικριτική ε, διανομή, ή ένα σύστημα επικριτική διανομή, δεν το αγγίζουν εδώ οι διατάξει που προτείνει η Κομισιόν. Οι κατασκευαστέ σαφώ μπορούν να συνεχίσουν να έχουν ένα σύστημα επιλεκτικής διανομή για να υπολάνε τα ανταλλακτικά του και τα εργαλεία του σε εξειδικευμένους αλλά εδώ λέμε ότι υπάρχει μια ανεξάρτητη αγορά για αγορά επισκευών και διαγνωστικά εργαλεία και το θέμα είναι το να υπάρχει ένα, μια ευρύτερη επικοινωνία των στοιχείων. Τώρα για την ασφάλεια των ανταλλητικών, κύριε Σβάμπ. Κρίμα που ο κύριος Χόλμκουιστ και δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για πληροφορίες για το θέμα της, του σχεδιασμού ανταλλακτικών ή σχέδια ή κατασκευή ανταλλακτικών. Η κλίπα, δημιουργούν, παράδειγμα, δημιουργούν ανταλλακτικά και για αγροτικά μηχανήματα και διασφαλίζουν ασφαλώς την ασφάλεια των ανταλλακτικών τους. Ε, ε, ε, τα, τα, οι αναρμονισμένες απαιτήσει εδώ πέρα ισχύουν. Αυτό για την ασφάλεια των ανταλλατικών. Αλλά επιπλέον εδώ συζητούμε για κάποιες πληροφορίες που θα πρέπει να είναι, ε, να είναι γνωστές για θέματα ασφαλείας. Και στον γύρο 5 και στον γύρο 6 αναφέρθηκαν τις συγκεκριμένες πληροφορίες συγκεκριμένες ε, για θέματα διατηρητικότητας. Δεν μιλάμε για σχέδια και κατασκευή ανταλλακτικών. Απλά μιλάμε για τον τρόπο που θα μπορούσαν οι ανεξάρτητοι επισκευαστές να, να εφαρμόσουν τα ανταλλακτικά στα οχήματα. Ε, το θέμα το να μην ε, μοιραζόμαστε τις πληροφορίες και να δημιουργούμε μια κλειστή αγορά έγινε αυτή η συζήτηση και στα εμπορικά οχήματα και στα βαρέα οχήματα παρόλο που υπάρχουν ε, εκεί πέρα ακόμα περισσότερα τεχνικά ζητήματα και εξειδικευμένα βρήκαμε τον τρόπο να κάνουμε τη μοίρα, να μοιραζόμαστε τι πληροφορίες. Λέτε ότι είστε διαφορετικοί από την αυτοκινητιστική βιομηχανία, αλλά μην το κάνετε λάθος. Τα εμπορικά οχήματα υπάρχουν πολλέ ομοιότητες και εμείς όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα λαμβάνουμε υπόψη αυτή τη στιγμή και καλό είναι να υπάρχει αυτό το μοίρασμα των πληροφοριών και δεν είναι απαραίτητο να είμαστε σε ένα δίκτυο, το δίκτυο των αντιπροσώπων, των dealer, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και ανεξάρτητοι επισκευαστέ. Αυτή θα δίνουν μια ελευθερία επιλογή και ε, κατά κλείδι οι τεχνικέ πληροφορίε θα πρέπει να είναι ε, ελεύθερα προσβάσιμε. Okay, ευχαριστώ όλους πολύ για την συνεισφορά σας και όλους τους ομιλητές. Θα καλέσω τώρα τον κύριο Ματινού να συνοψίσει και θα δώσω και το λόγο στον κύριο Παντζέρη για να ολοκληρώσουμε την ακρόαση. Θέλετε να πείτε κάτι τώρα? Ε, μιλήστε, δεν είχατε δυνατότητα πριν. Άφησα την γειτόνισά μου να μιλήσει και να κάνει την πρότασή της απλώς σχετικά με αυτά που υπόθηκαν και αυτά που αναφέρθηκαν. Από ό,τι γνωρίζω κάνετε διάφορες εξτατείες στις χώρες της Ενώσης και λέτε ότι δεν ε, βλέπουμε ανεξάρτητα δίχτυα επισκευαστών. Είναι για λόγους μη τεχνολογικούς, διότι η διάδοση των πληροφοριών δεν σημαίνει αρμοδιότητα στην, της χρήσεως. Είναι πολύ περίπλοκο να, αποκτήσει κανείς αυτή την, ε, την άδεια και συνδέεται με το δίκτυο των κατασκευαστών. Είναι μικρή η αγορά, οι δεξιότητες και λοιπά και οι γνώσεις. Λέτε είναι μικρή αγορά, εφαρμόζουν τι συνταγέ. Αλλά ο άνθρωπο είναι εκείνο που πρέπει να εφαρμόσει την τεχνική. Και υπάρχουν λίγοι τεχνικοί καταρτισμένοι, αρμόδιοι, ικανοί για να το κάνουν αυτό. Ε, και κάποιο άλλο το είπε αυτό. Είναι πρόβλημα ανταγωνισμού. Τα δίκτυα ανταγωνίζονται το ένα το άλλο, ηρίστον παρόδο. Και αλλάζουν ε, διανομή στα δίκτυα. Δεν είναι κάτι σταθερό και αντιπροσώπους. Αλλά ο ανταγωνισμό δεν είναι κατάσταση το είπατε αυτό. Διότι αληθεύει ότι στην επαγγελματική πρακτική διαπιστώνω, διαπιστώνεται μάλλον στη Γαλλία, ότι πολλοί εμπειρογνώμονε από τον τομέα των αυτοκινήτων ασχολούνται με τα αγροτικά, ε, ασχολούνται με αγροτικά θέματα από την έποψη των αυτοκινήτων και οδηγούνται σε επικίνδυνε λύσεις για την ασφάλεια των ατόμων. Υπάρχουν ίσως προβλήματα ανταγωνισμού και ίσως προβλήματα ασφαλείας, αλλά τα δύο δεν είναι αλληλένδετα. Αποκάλυψη πληροφοριών, πρόσβαση στι πληροφορίε. ποτέ δεν θα βοηθήσει κάποιον ο οποίο δεν έχει τις δεξιότητες αν δεν έχει την κατάρτιση διαρκείας, γιατί χρειάζεται διαρκή κατάρτιση. Δεν είναι απλώ ένα σασί, τέσσερι τροχοί και ένα κινητήρα. Είναι πολύ περισσότερο από όλα αυτά. Right. Well, thank you very much. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι δευτερολόγησαν. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ματινόφ. Να σας δώσω τέσσερα λεπτά για να ανακεφαλαιώσετε. Κάτι αναφέρθηκε πριν. Δεν ξέρω αν καλύψατε την πρόταση τη ΣΥΜΑ που εγκρίθηκε και από άλλους. Να υπάρχει διτή ε, κατηγοριοποίηση για τα τρακτέρ ε, υψηλής ταχύτητας και χαμηλής ταχύτητας, ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή δομή, ξεχωριστή πρόβλεψη αποκλειστική για τα τρακτέρ ε, υψηλής ταχύτητας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μιλάμε για θέματα ασφάλειας και περιβαλλοντικά. Δεν θα μιλήσω μόνο για τις πληροφορίες, για τις επισκευές και συντήρηση, με μία εξαίρεση, γιατί δεν θα αντισταθώ εντελώς στον πειρασμό. Να ευχαριστήσω και εσάς που οργανώσατε τη συζήτηση αυτή. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και επιβεβαιώνω ότι από άποψη κομισιών εμεί συνεργαστήκαμε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά μαζί σας για θέματα ασφάλειας και περιβαλλοντικά θέματα. Είμαι ευγνώμων που μας θυμήσατε ότι δεν είναι αυτοκίνητα οι ελκυστήρες. Αυτό εμείς το παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, αν θέλετε, αυτής της νομοθεσίας. Ειδικά διότι επιπροσθέτως αποκλείομαι από την οδηγία για τα μηχανήματα του ελκυστήρες και πρέπει να φροντίσουμε όλα τα στοιχεία και ειδικότερα τα θέματα ασφάλειας θα πρέπει να λαμβάνονται παρκώς υπόψη να θυμίσω ότι ο στόχος της συγκεκριμένης πρότασης είναι να θέσει ένα πλαίσιο που θα συμπληρωθεί με από συγκεκριμένες κατεξουσιοδότηση πράξεις που θα αναφέρονται συγκεκριμένα στις απαιτήσεις. Ένα σύστημα που θα επιτρέψει με την ε, απαραίτητη μεθοδολογία τα επόμενα χρόνια να προσαρμόζεται όχι μόνο στην τεχνολογική ανάπτυξη, εξέλιξη, αλλά θα λαμβάνει υπόψη και πρόσθετες ανάγκες ενδεχομένως για την καλύτερη ασφάλεια και το, την προστασία του περιβάλλοντος. Θα προσαρμόζεται το σύστημα δηλαδή για να ενσωματώνει νέες απαιτήσει ή να προσαρμόζει τις υφιστάμενες. Αυτή είναι η ουσία του. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κάτι τέτοιο. την Κυριακή κοίταγα τις εφημερίδες στην Ιταλία και υπήρχε ένα ενδιαφέρον άρθρο για τα ατυχήματα με τους ελκυστήρες Βέβαια οι στατιστικές ε, δεν είναι τέλειες, αλλά αν δούμε ας πούμε το 2010 τα στοιχεία ήταν 38,3% περισσότερα τα ατυχήματα από πέρσι. Η ασφάλεια λοιπόν είναι θέμα οπωσδήποτε. Πρέπει να φροντίσουμε όπως τα ακούσαμε ότι ό,τι και να ε, φροντίζομαι στα πλαίσια της οδηγίας για τα μηχανήματα να το ε, λύνουμε και στην νομοθεσία για τα τρακτέρ και στην ε, μεθοδολογία εργασίας μας έχουμε και την ε, ε, κανονιστική επιτροπή, έχουμε και ομάδα εργασίας όμως και θα έχουμε και μια άτυπη ομάδα εργασίας για θέματα ασφάλειας κατά την εργασία, γιατί ανάμεσα στα διάφορα θέματα ασφαλείας και αυτό είναι πολύ κύριο ζήτημα. Τέλος, η πληροφορία για στα πλαίσια επισκευών και συντήρησης. Το μήνυμα είναι, αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχουν οι βασικές αρχές στην νομοθεσία και είμαστε ανοιχτοί για να ορίσουμε με ακριβή και στοχευμένο τρόπο τα μέτρα στην πράξη κατά εξουσιοδότηση. Γνωρίζομαι τις ιδιαιτερότητες του τομέα των ελκυστήρων. Δεν θα αντιγράψουμε τις διατάξεις ε, από τα επιβατικά και τη σχετική νομοθεσία. Ξέρουμε ότι πρέπει να το δούμε προσεκτικά το θέμα αυτό, που είναι σημαντικό όμως, είναι η αρχή. Και πάλι δεν μπορώ να αντισταθώ, σα το είπα κύριε Πρόεδρε, ε, δεν μπορώ να αντισταθώ να μιλήσω για τη νομική βάση. Η ίδια νομική βάση που είναι το πρώην άρθρο 95 και τώρα είναι το 114 της συνθήκης, έχει χρησιμοποιηθεί για διάφορους ε, κανονισμούς ε, έγκρισης τύπου χωρίς ε, να έχει αμφισβητηθεί η νομική βάση και η υποχρέωση πρόσβασης σε πληροφορίες συντήρησης επισκευαστής είναι ενσωματωμένη στη διαδικασία έγκρισης τύπου. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε λοιπόν σε θέματα πολιτικής Νομοθεσία ανταγωνισμού. Όλα αυτά τα στοιχεία τα εξετάζουμε πολύ με την νομική υπηρεσία και του συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Ούτε έχουμε πρόθεση να πειράξουμε το παρόν σύστημα διανομής και του συσχετισμού του. Αλλά η αρχή πρέπει να διατηρηθεί και να ορίσουμε πολύ στοχευμένα μέτρα στην κατεξουσιοδότηση πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ματίνο που παρενέβητε δύο φορές και σχολιάσατε ορισμένα από τα θέματά μας. Πολύ δουλειά μένει να γίνει ακόμη και ο κύριος Παντσέρη έχει να σκεφτεί πολλά έχοντας ακούσει αυτά που άκουσε σήμερα. Έχει την θέση ως εισηγητής και τώρα θα του δώσω την ευκαιρία να συνοψίσει τη συζήτηση και να μας μιλήσει για το μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών καθώς ε, προχωρούμε στο τελευταία φάση εξέταση αυτής της σημαντικής πρότασης. Κύριε Σπαντσέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τη διαθεσιμότητα που δείχνετε να το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ όλους σας για τις συνεισφορές σας που είναι χρησιμότατες για τη σύνταξη της εκθέσεως. Μπορώ να πω συνοπτικά, εξαιρετικά συνοπτικά το εξής. Υπάρχει επίγνωση της σημασίας που έχει ο τομέας και την απέτηση που υπάρχει να θεσπιστεί ένας κανονισμός που μέσω πλέον εναρμονισμένων διατάξεων θα μπορεί να εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν το σκοπό είναι καλό να προχωρήσουμε αυτήν την απόψή μας, να μην ε, αλλάξουμε την τοποθέτηση, αλλά να κάνουμε κάποιες τροποποίησεις οι οποίες να ταιριάζουν με το γενικό στόχο για τα διάφορα σημεία. Εκφράζει την άποψή μου τώρα. Προς τα ποια κατεύθυνση να κινηθούμε, ποια γραμμή να ακολουθήσουμε. Σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δούμε τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, ποιους δρόμους, τι θα πρέπει να εισάγουμε. Χρονοδιάγραμμα, Κατάλαβα αυτά που υπόθηκαν. Υπάρχει πρόβλημα υπερφόρτωσης νομοθετικής. Προσφάτως έγιναν διάφορες παρεμβάσεις, προβλέφθηκαν διάφορες παρεμβάσεις και πριν φτάσουμε στον εφησυχασμό για να εφαρμοστεί ο κανονισμό του 1η του 2014, να μην ξεκινήσουμε από το 0 με πλήρη μία, να αξιολογήσουμε αν υπάρχουν περιθώρια για να πάρουμε να συμφωνήσουμε μια μετάθεση σε εφαρμογή του κανονισμού ή αν σεβόμενοι τις προθεσμίες μπορούμε σταδιακά να εφαρμόσουμε τον κανονισμό. Δύο ενδεχόμενα. Μπορούμε να τα εξεργαστούμε. Θα δω τι περιθώρια λιγμών υπάρχουν για να πετύχουμε το στόχο μας. Για το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε μέχρι πρόσφατα, πρόσφαση στις τεχνικές πληροφορίες. Κατανοώ άριστα τα προβλήματα που έχουν κάποιες επιχειρήσεις όσον αφορά τις πληροφορίες. Θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα εγγυήσεων που θα δημιουργηθεί έτσι θα μπορούμε να ανταποκριθούμε σε απαιτήσει των επιχειρήσεων, αλλά και σε εκείνες στους επισκευαστές, εκείνους που πολλούν τα ανταλλακτικά και τους χρήστες. Όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το θεωρώ σημαντικότατο το κεφάλαιο αυτό, διότι διασυνδέεται και με την ασφάλεια. Και την οδική ασφάλεια, αλλά και των εργαζομένων Πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Πρέπει να συμβιώσουν και οι αντιπρόσωποι και οι επισκευαστές που συνδέονται με την κατασκευαστική εταιρεία και οι ανεξάρτητοι να συμβιώσουν. Για να αποφύγουμε και διαταράξεις και να μην δημιουργήσουμε στρεβλώς στην αγορά. Χρειάζεται σοβαρή αξιολόγηση. Μετά από αυτά που άκουσα για το κεφάλαιο 16 θα έλεγα προσωπικά ότι αν παραμείνει έτσι μπορούμε να το βελτιώσουμε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το κεφάλαιο 16. Μπορούμε να επεξεργαστούμε μια βελτίωση του κειμένου. Μετά ετέθη το θέμα της ασφάλειας. Χρειάζεται εμβάθυνση εδώ πιστεύω. Κάποια εμβάθυνση. Και επί τη βάση της πρόσφατης ανάγνωση αυτό που είπατε για αυτά που έγραφε μια Ιταλική εφημερίδα. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουν περισσότερες απαντήσεις σε αυτό το τομέα, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις πληροφορίες που συμπεριλαμβάνουν. Δεν ξέρω αν θα είναι εφικτό αυτό. Πρέπει να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσουμε ίσως και ένα δίκτυο φορέων που μπορούμε να συμβολευτούμε ε, για να πετύχουμε τους στόχους θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο, δεν είναι κακή ιδέα. Θα μπορούσε να αναφερθεί και στον κανονισμό. Τέλος, δύο πράγματα. Για τα κινητά μηχανήματα. Όλοι πιστεύουν ότι χρειάζεται να ρυθμιστεί το κεφάλαιο. Κάποιος λέει να βγει εκτός, κάποιος όχι εκτός. Εγώ θα έλεγα να μην βγάλουμε το κεφάλι αυτό τον κανονισμό. Να δούμε μπορεί να υπάρξει ένα δεδειγμένο παράτημα που θα καλύπτει αυτή την περίπτωση και να ταιριάζει με τον υπόλοιπο κανονισμό η προσέγγιση. Τα side by side και τα ATV e ε, μπορούσε να βγει μια νέα κατηγορία T6 σύμφωνα με αυτά που άκουσα. Με έπεισαν αυτά που άκουσα. Είναι νέο παιδί όμως και χρειάζεται εμβάθυνση ο προβληματισμός. Να σε ευχαριστήσω εκ νέου για τη συμμετοχή σας, για την συμβολή σας. Μετά από αυτή την ακρόση, Έχουμε συζήτηση όσον αφορά το σχέδιο εκθέσεως στις 24, μάλλον 14 και 16 Ιουνίου, μετά προθεσμία για τις τροπολογίες 6 Ιουλίου, συζήτηση επί των τροπολογιών 4 με 6 Οκτωβρίου, ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ περίπου 17 Οκτωβρίου και στην Ολομέλεια Νοέμβριο φέτος. Έχουμε τον αναγκαίο χρόνο, ούτω ώστε αυτά που έθελαν συζήτηση να ληφθούν υπόψη στην έκθεση που θα πρέπει να συνταχθεί. Με τη συνεισφορά όλων των σκιωδών εισηγητών βεβαίως που ήταν εδώ παρόντες. Και κυρίως ε, να θα αναλυθεί υπόψη η συνεισφορά του Προέδρου. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο, Ευχαριστώ, κύριε Παντζέρη. Αυτά τα θόρμητα χειροκροτήματα δείχνουν την εκτίμηση στο πρόσωπό σας. Και ευχαριστούμε και όλους τους ε, εμπειρογνώμων που μίλησαν εκ μέρους Επιτροπής. Υπάρχει και το Συμβούλιο που είναι συνεταίρο μα στη συναπόφαση. Το Συμβούλιο επεξεργάζει την οδηγία για του ελκυστήρε. Περίπου Οκτώβριο-Νοέμβριο θα καταλήξουν σε συμπεράσματα. Γι' αυτό παρατείναμε το χρονοδιάγραμμα. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τις συζητήσεις στο, στο Συμβούλιο. Ελπίζουμε να συμμετάσχει περισσότερο στις συζητήσεις και το Συμβούλιο και να συνεργαστεί μαζί μας. Δεν με απομένει παρά να κηρύξω τη λήξη συνεδρία σα. Ευχαριστώ όσου παρακολουθούν από την ιστοσελίδα μα. Έχουμε και το, το έντυπό μας εδώ, το newsletter, το πιο πρόσφατο ε, έντυπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, στείλτε μας ένα email, να σας στείλουμε μέσω διαδικτύου το έντυπο και όποιος από τους ομιλητές θέλει να γίνει φίλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς μπορεί να υπογράψει, να γίνει μέλος και θα σας ενημερώνουμε για την οδηγία περί ελκυστήρων καθώς και ε, τα μέτρα για, τους, για τις μοτοσυκλέτες και για τα άλλα προγράμματα που έχουμε μπροστά μας. Σας ενημερώνουμε μέσω του newsletter. Σας καλούμε να είστε φίλοι της Επιτροπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξανασυνεδριάσουμε αύριο το πρωί στις 9. Έχουμε πληρέστατη μερίσια διάταξη. Ψηφίζουμε στις 10 επί διαφόρων γνωμοδοτήσεων. Λίγη σημερινή μας συνεδρίαση και σας περιμένω, σας δω αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα.